So, good morning, dear colleagues. Καλημέρα αγαπητοί συνάδελφοι. Με χαρά καλωσορίζω τον Αντιπρόεδρο Ντομπρόφσκη. Είναι η πρώτη του εμφάνιση αυτή τη χρονιά στην ε, Επιτροπή μας. Είναι για τις κεφάλαια αγορές και την Ένωση κεφαλαία και την οικονομική σταθερότητα ε, φυσικά τα λέμε πολύ συχνά. Σήμερα θα εστιάσουμε στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, την Τραπεζική Ένωση, την ε, Ένωση Κεφαλαίου Αγορών. Η Επιτροπή έχει κάνει πολλές νέες προτάσεις για νομοθεσία σε αυτό τομέα ιδιαίτερα για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, τα επενδυτικά ταμεία και τις διαμεθοριακές αμοιβέ και άλλα. Όπως ξέρετε, η Επιτροπή στοχεύει να παρουσιάσει την επόμενη εβδομάδα σημαντικές προτάσεις. Και εμείς πιέζουμε για περισσότερη πρόοδο στην Τραπεζική Ένωση. Πρώτα απ' όλα για του κανόνε, για το πακέτο μείωση των κινδύνων, το λεγόμενο, και για την ολοκλήρωση τη Ευρωπαϊκή Ένωση, το πρόγραμμα εγγύηση των καταθέσεων. Πρέπει να εκφράσω την ανησυχία μου, διότι στο Συμβούλιο, αλλά και εδώ, δεν φαίνεται να είμαστε σε θέση να προωθήσουμε από κοινού ορισμένα θέματα και παράλληλα. Και αυτό μας ανησυχεί, γιατί εγώ θέλω να υπάρξει προώθηση και του προγράμματος για τη μείωση των κινδύνων για την Ένωση Αγορών και γενικά τις ε, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Υπάρχει κάποια πρόοδος. Χθες έγιναν δύο πολύ σημαντικέ ψηφοφορίες για την αναδιατύπωση του ΕΜΙΡ και το ΕΜΙΡ 2 και για τις εταιρείε επενδύσεων προχωράμε. Ε, εργαζόμαστε και για την αναθεώρηση του ΕΣΑ. Άρα το Κοινοβούλιο θέλει να προωθήσει για όλα αυτά τα θέματα που είναι τόσο στενά άλληλο συνδεδεμένα. Αλλά, κύριε Επίτροπε, παρακαλώ, να σας δώσω το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, καταρχάς σας ευχαριστώ για αυτή την πρόσκληση να συζητήσουμε το κοινό μας έργο για, μια, για πιο ανθεκτικό και ολοκληρωμένο χρηματοστατικό τομέα στην Ευρώπη. Όπως η ερηνή πρόβλεψη Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρόσφατα βεβαίως, η οικονομία μας αναπτύσσεται με τους ταχύτερους ρυθμούς που είχε για μια δεκαετία ταυτόχρονα. Η πρόβλεψη μας έδειξε κινδύνους όσον αφορά την οικονομική ανάπτυξη να ελοχεύουν, αυξανόμενο προστατευτισμό και γεωπολιτικές ε, εντάσεις. Αυτό σημαίνει ότι το παρούσα το περιθώριο ευκαιρίων περιορίζεται. Θα πρέπει να συμφωνήσουμε σύντομα πώς να δημιουργήσουμε σκληρά θεμέλια για την Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Βασικό τμήμα αυτών των εργασιών είναι η ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης και να δημιουργήσουμε τα ε, τα βασικά εργαλεία για την ε, Ένωση των Κεφαλαιογορών. Λοιπόν, αυτά θα είναι τα δύο πρώτα μου θέματα για σήμερα. Ταυτόχρονα, τώρα είμαστε σε μια καλή θέση, ούτως ώστε να μπορούμε να κοιτάξουμε προ μελλοντικέ ευκαιρίε και δυνατότητε. Πιο συγκεκριμένα θέλουμε ο χρηματοστικός τομέας της Ευρώπης να ηγηθεί στον κόσμο όσον αφορά τα βιώσιμη χρηματοπιστωτική προσέγγιση και έχουμε αντικοποίησει αυτή την άνοιξη τη προσπάθεια στον τομέα. Και αυτό θα είναι το τρίτο θέμα μου σήμερα. Θα ξεκινήσω από την Τραπεζική Ένωση. Η πρόσφατη ετήσια έκθεση όσον αφορά την Τραπεζική Ένωση ε, από το Σάντερ Λούνς έδειξε ότι έχουμε, κάνει, έχουμε πετύχει βελτιώσει όσον αφορά το ρυθμιστικό και υποπτικό πλαίσιο για τις τράπεζες αλλά διαχειριστούμε μια τραπεζική κρίση με το λιγότερο αντίκτυπο για τη χρηματοδοτική σταθερότητα και σωρολογούμενους θα πρέπει να ολοκληρώσουμε το παρόν σύστημα. Η προσέγγιση μας αποφασίζεται στη μείωση του κινδύνου και τον επιμερισμό του κινδύνου. Αυτά πηγαίνουν μαζί. Το πρώτο βήμα θα πρέπει να είναι να καταλήξουν τελικά σε συμφωνία στο πακέτο για τις τράπεζες του Νευρίου 2016 για να μειώσουν περαιτέρω τους κινδύνους στο τραπεζικό τομέα. Ελπίζω ότι παρόμοιο έργο εδώ στο Κοινοβούλιο θα ολοκληρωθεί σύντομα ε, με τον Γκούναρ Χόκμαρ και τον Πίτερ Σάιμον. Είναι πολύ σημαντικό ο χρόνο, διότι αν έχουμε και άλλε καθυστερήσει, ίσω υπονομεύσουμε το στόχο μα να πετύχουν πολιτική συμφωνία πριν τι εκλογέ του επομένου έτου. Λοιπόν, κινόμαστε ένα ε, κοινό σταθμό για, την, για το ενιαίο σύστημα καθάρισης. Θα πρέπει να ενισχύσουμε την πιστοσύνη στο τραπεζικό σύστημα και θα πρέπει ε, να μειώσουμε τους κινδύνους. Χρειαζόμαστε σαφήνεια όσον αφορά το σύστημα το ευρωπαϊκό για την ε, ασφάλεια των καταθέσεων και προσλέπω στο έργο του Έστερ Ντελάγκε και του σχεδόν εισηγητών για να αναπτύξουμε συμβιβαστικέ. Τον Μάρτιο υφετήσαμε ένα πακέτο για τα για τα κόκκινα δάνεια είναι ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους για το τραπεζικό σύστημα στην Ευρώπη σήμερα. Ακόμα και αν έχει μειωθεί ο κίνδυνος μετά την κρίση, το πακέτο συμπεριλαμβάνει διάφορα πακέτα να βοηθήσουμε τις τράπεζες να επεξεργαστούν τα υψηλά επίπεδα των κόκκινων δανείων και να παρεμποδίσουν μια τέτοια σώρευση στο μέλλον. Ελπίζω ότι το έργο του ουσιαστικό επί των προτάσεων σύντομα θα ξεκινήσει στην Επιτροπή σας και τώρα ας προχωρήσω και να πάω στην Ένωση των Κεφαλαγορών. Μαζί ήδη έχουμε πετύχει πολλά όσον αφορά τα κεφάλαια κινδύνου, ε, τα εγχειρίδια και την ασφάλεια αυτών των επενδύσεων, αλλά από 13 νομοθετικέ προτάσει που βλήθησαν μέχρι τώρα, οι 10 ακόμα τελούν εν αναμονή για υιοθέτηση από του συνομοθέτε. Λοιπόν, πρέπει να επιταχύνουμε το έργο μα, ούτω ώστε αυτέ οι προτάσει να περάσουν τη γραμμή του τερματισμού πριν από τι επικείμενε ευρωπαϊκέ εκλογέ. Ε, ε, ταχύτατα θα έχουμε την ε, απόσυση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ενιαία αγορά και αυτό αυξάνει τον καταπικό χαρακτήρα του θέματος. Θα ήθελα να ειστεστείτε επί τριών βασικών διαστάσεων της ενώσεως των κεφαλαγορών Πρώτα απ' όλα θέλουμε οι καταναλωτές και οι επενδυτές να ωφεληθούν πλήρως από την ενιαία αγορά χάρη ε, σε διάφορα χρηματοδοτικά προϊόντα που καλύπτουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα σημαντικό παράδειγμα ήταν η πρόταση του περασμένου Ιουνίου για πανευρωπαϊκό προϊόν για τη συντάξιση, το ΠΕΠ. Ευχαριστώ την εισηγήτρια Σοφίν Τεβέλτ και τους κύριους εισηγητές για τις προσπάθειες μέχρι τώρα και ε, βασίζομαι ότι θα έχω θέση τη Επιτροπή στο χαρτοφυλάκιο πριν τι θερινέ διακοπέ. Πριν από δύο μήνε παρουσιάσαμε αρκετέ προτάσει για να προωθήσουμε διάφορα προϊόντα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω μια άδεια τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω για συλλογή πόρων μέσω crowdfunding και διάφορα μέτρα να μειώσουμε ε, κανόνες για, ε, για τα ομόλογα που καλύπτονται και να μειώσουμε του φραγμούς για συνοριακή κατανομή των επενδυτικών πόρων. Θα πρέπει όλοι οι Ευρωπαίοι να μπορούν να κάνουν συνολικέ πληρωμέ ευρώ για στην ίδια τιμή όπω και στο εσωτερικό τη χώρα του. Στόχο είναι να θετήσουμε κάθε μία από τι προτάσει εντό ε, τη παρούση θητεία και ελπίζω ότι θα τύχω τη υποστήριξή σα και να ξεκινήσουν οι εργασίε πάρα πολύ γρήγορα και πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τα χαρά να παράσχουμε οποιαδήποτε αρρωγή που απαιτείται. Την επόμενη εβδομάδα θα στηρίξουμε αυτό το κατάλογο νομοθετικών προτάσεων, ούτω ώστε να μπορέσουμε ε, τα κρατικά ομόλογα να τα υποστηρίξουμε και τους διάφορους κρατικούς τίτλους, η SBBS. Αυτό θα βοηθήσει περαιτέρω ολοκλήρωση και επικοινομορφία εντός του χρηματοδοτικού τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα βοηθήσει ε, να μειωθούν οι διάφοροι κίνδυνοι από τα κρατικά χρέη των τραπεζών. Αυτοί οι τίτλοι θα εκδίδονται από συμμετέχοντες στην αγορά και οπότε δεν θα υπάρχει επιμερισμός ε, και διάδοση των κινδύνων και των απολειών και η πρότασή μας δεν θα συνεπάγεται ε, διάφορες αλλαγές όσον αφορά τα διάφορα μέσα για την αντιμετώπιση των κρατικών χρεών. Η δεύτερη διάσταση εστιάζεται σε περισσότερη, καλύτερη υποπτία των κεφαλαιογορών τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω, ώστε οι κανόνε να εναρμονιστούν στην πράξη και να μην είναι απλώ άσκηση επιχάρτου. Λοιπόν, θα ήθελα εδώ να συγχαρώ την Τανούτα Χούμπνερ για την ε, ομαλή υιοθέτηση της εκθέσεως όσον αφορά την πρότασή μα να ενισχυθεί η υποπτία των ε, κεντρικών ε, συμβαλωμένων μερών είναι ένα καλό παράδειγμα αυτό που δίνει το Κοινοβούλιο και θα πρέπει να προωθήσει τα κρατη μέλη συμβαστούν και βασίζομαι στο Κοινοβούλιο να ηγηθεί και σε άλλα χαρτοφυλάκια τώρα που πλησιάζουν προς το τέλος της θητείας. Ε, ταυτόχρονα τεθήθηκε εδώ και η έκθεση Wenden Langer για την αδιατύπωση του Εμμύρ, για το Refit και το Εμμύρ. Και νωρίτερα αυτό το έτος ε, ενεκρίθη η έκθεση Case Winburn και Jacob von Weizsäckers για την ανάκτηση του CCP και την επίλυση των διαφόρων προβλημάτων. Θα ήθελα να ευχαριστήσω του για το έργο του. Θα πρέπει να διατηρηθεί αυτή η ορμή όταν εξετάσουμε τον εποπτικό συντονισμό σε άλλου τομεί, όπω και όσον αφορά την πρότασή μα για την αναθεώρηση της λειτουργία ε, των ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών. Πρέπει να, να εξοπλίσουμε καλύτερα αυτού του εποπτικού φορεί για να υπάρχει καλύτερη σύγκληση και να αντιμετωπιστούν νέε προκλήσει. Το Κοινοβούλιο ε, σημείωσε το ίδιο πόσο σημαντικό είναι αυτό το θέμα για να στηριχθεί ε, η ανάπτυξη τη ε, Ένωση των Κεφαλαγορών. Προσβλέπω στο σχέδιο εκθέσεώ σα και βασίζομαι στου συνεισηγητέ να τηρήσουν το σχεδιασμένο χρονοδιάγραμμα, ώστε να πετύχουμε μια συμφωνία τον επόμενο χρόνο. Τώρα έρχομαι στο τρίτο σημείο, δηλαδή να αρθούν οι φραγμοί για την εμβάθυνση των κεφαλαγορών και να υπάρχουν σαφέστεροι και απλούστεροι κανόνες για τις εταιρείε. Ε, με την αίτησή μα να δοθούν στοιχεία εντοπίσαμε μέτρα για την απλούστερη των κανόνων και να μειωθεί το διοικητικό άχθο για τι εταιρείε και έκτοτε αυτό αποτελούσε ε, προτεραιότητα ε, για την επόμενη επίσης ε, νομοθεσία. Τον επόμενη εβδομάδα θα προτείνουμε πιο ανάλογους κανόνες για να μπορούν να κατατάσσονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι η ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας και η Ένωση των Κεφαλαγορών της Ένωσης δεν μπορεί να οικοδομηθεί χωρίς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και τώρα πάω στο τρίτο τελικό σημείο τη εισαγωγική μου παρέμβαση για τη σημαντική νέα ευκαιρία που έχει ο χρηματοστατικό μα τομέα, δηλαδή η ε, βιώσιμη και πράσινη χρηματοδότηση και σχετικό μέσο είναι σημαντικό για πολλού λόγου, διότι η χρηματοδοτική σταθερότητα εν ώψη των καταστροφικών συνεπειών τη αλλαγή του κλίματο είναι κάτι πολύ σημαντικό. Από το 2007 μέχρι το 2016, οι οικονομικέ απώλειε από ε, καταστροφέ λόγω καιρού αυξήθηκε κατά 86%. Λοιπόν, καλωσορίζω την υποστήριξη του Κοινοβουλίου για πολλέ από τι δράσει από αυτού του θέματο, όπω εκφράζεται στην έκθεση Ιδέα Πρωτοβουλία τη Μόλι Σκοτ Κάτω. Την επόμενη εβδομάδα θα παρουσιάσουμε την πρώτη ομάδα των τεσσάρων προτάσεών μας. Πρώτα θα ξεκινήσουμε τη διαδικασία σχεδιασμού συστήματος ταξινόμησης για την Ευρωπαϊκή Ένωση για βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες. Αυτό θα βοηθήσει επίσης να καθορίσουμε κριτήρια για μελλοντικά πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και ε, κατονομασία για κρίσινα χρηστοτικά προϊόντα όπως είναι τα πράσινα ομόλογα και επενδυτικά ταμεία. Ε, δεύτερον θα προ τίνουμε την περιγραφή του πώς, μπορούν, πώς αυτοί που χειρίζονται επενδύσεις εκ μέρους άλλων θα πρέπει να αποκαλύπτουν το πώς ενσωματώνουν τη βεσιμότητα στις διαδικασίες τους Τρίτον, θα προτείνουμε τη δημιουργία νέων κατηγοριών βαθμολόγηση που θα δίνει περισσότερε πληροφορίε στου επενδυτέ όσον αφορά ε, τα διάφορα, το ίχνο άνθρακο για διάφορα χατοφυλάκια. Τελικά, θα προτείνουμε το ότι οι επενδυτικέ εταιρείε και οι ασφαλιστέ θα πρέπει να εξετάζουν τι προτιμήσει βιωσιμότητα κάθε πελάτη όταν δίνουν συμβουλέ για επενδύσει. Το σχέδιο δράση για ε, βιώσιμη χρηματοδότηση του Μαρτίου φέτο συμπεριλαμβάνει περαιτέρω έξι δράσει που θα δρομολογηθούν από τώρα μέχρι το τέλο αυτή τη θητεία. Πιο συγκεκριμένα, υποστηρίζουμε τις προτάσεις του Πίτερ Σάιμον για πράσινο υποστηρικτοϊκό παράγοντα για να προωθηθούν τα πράσινα δάνεια και επενδύσεις και καλύτερη συμπερίληψη της βιωσιμότητα στη διαχείριση κινδύνου των τραπεζών και είμαστε έτοιμοι να παράσχουμε όλη την αναγκαία υποστήριξη για να εντοπιστούν ε, τα, οι πιο ορθοί προληπτικοί τρόποι για να εφαρμόσουμε αυτούς, αυτές τις προτάσεις. Λοιπόν, αξιότιμα μέλη, Τώρα είμαστε μόλις ένα έτος πριν από τις επόμενες εκλογές για το Ευρωκοινοβούλιο. Λοιπόν, ας αδράξουμε αυτή τη στιγμή, ας την εγκαταλευτούμε, ας δραστηριοποιηθούμε τώρα. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό, να ολοκληρώσουμε αυτό που ξεκινήσουμε όσον αφορά την Τραπεζική Ένωση και την Ένωση των Κεφαλαγορών και έτσι μπορούμε να καταστήσουμε τις οικονομίες μας και τον χρηματοδοτικό μας τομέα πιο ανθεκτικούς ε, και να προσαρμοσμένους για το μέλλον. Ελπασίζομαι λοιπόν και ελπίζω ότι θα έχω την υποστήριξή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε, κύριε Αντιπρόεδρε της Επιτροπής, για την ευρεία και ολοκληρωμένη παρουσίαση των θεμάτων και πρωτοβουλειών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και για την έκκλησή σας για να υπάρξει υπεύθυνη δράση. Αυτό είναι αναγκαίο και το χαιρετίζουμε. Ελπίζω το Κοινοβούλιο να ανταποκριθεί σε αυτές τις προκλήσεις, να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων. Για να καταλήξουμε σε όλα αυτά τα νομοθετικά θέματα που έχουν ευρίες και άλλο συνδεδεμένες επιπτώσεις. Και για να ολοκληρωθεί η προσπάθειά μας ε, χρειάζονται όλα αυτά τα βήματα. Και ελπίζω και η διαπραγματευτική ομάδα για τα θέματα CRA, CRD να λάβει υπόψη αυτές τις εκκλήσεις. Γιατί θέσατε τόσο πολλά θέματα που είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε και μια πολύ καρποφόρα και ζωηρή συζήτηση. Ο κύριος Μπούρχαρτ Μπάλτς είναι ο πρώτος ομιλητής. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ και κύριε Ντομπρόφσκης που είστε παρόν σήμερα για αυτόν τον ε, διαρθρωμένο διάλογο. Φυσικά εκτιμώ το ότι αναφερθήκατε σε όλα τα σημαντικά θέματα. Αλλά όπως ε, σωστά είπατε, φτάνουμε στο τέλος της ε, θητείας. Αλλά τα θέματα που μας έχετε υποβάλει θα μας πιέσουν πολύ στο επόμενο χρονικό διάστημα. Δεν έχουμε αρχίσει τη συζήτηση 20 νομοθετικών θεμάτων. Και αυτό δεν συμπεριλαμβάνει και τις εκκρεμούσες προτάσεις που ακόμη ε, θα μας υποβάλλεται. Για παράδειγμα τα θέματα διακυβέρνησης, FinTech και το πρόγραμμα δράσης για την βιώσιμη χρηματοδότηση. Ελπίζω να συμφωνείτε ότι δεν μας αφήνεται καμία άλλη δυνατότητα παρά να ιεραρχήσουμε κάποια θέματα και Δηλαδή να κάνουν μια εράρχηση και να δώσουν προτεραιότητα σε κάποια θέματα. Λοιπόν, η ερώτησή μου, κατά συνέπεια, εσείς που είστε ο υπεύθυνος αντιπρόεδρος και επίτροπος, ποια θέματα για σας έχουν την υψηλότερη προτεραιότητα. Ποια θέματα θα θέλατε και αναμένετε να καταλήξουν κατά αυτήν τη θητεία. Έχω και άλλες ερωτήσεις, αλλά θα αρκεστώ σε αυτό για να έχετε περισσότερο χρόνο για τις απαντήσεις σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, ξέρετε ότι εγώ ε, πιστεύω ότι μπορούμε να καταλήξουμε για όλα αυτά τα θέματα. Είναι δυνατόν, είναι δυνατόν. Αυτό που κάναμε στο CCP, για παράδειγμα, δείχνει ότι ακόμη και ένα πολύ περίπλοκο και βέστο θέμα μπορεί να αντιμετωπιστεί. Εν πάση περιπτώσει, εσεί κύριε Επίτροπε, τι λέτε από αυτόν. Και εγώ συμμερίζομαι την ε, φιλοδοξία του Προέδρου Καλτιέρη να καταλήξουμε για όλα αυτά τα θέματα. Αυτή θα ήταν η ιδεώδης κατάσταση. Αυτό θα θέλαμε να επιτύχουμε. Αν βέβαια πρέπει να γίνουν κάποιες ε, επιλογές, είμαστε σε δύσκολη θέση γιατί όλες αυτές οι προτάσεις ε, πρέπει να προωθηθούν. Τις υποβάλαμε γιατί υπήρχε ανάγκη. Πιστεύω ότι πρέπει να στοχεύσουμε κυρίως να ολοκληρωθούν θέματα που εκκρεμούν εδώ και πολύ καιρό. Ολοκλήρωση του τραπεζικού πακέτου θα έλεγα. Οπωσδήποτε είναι σημαντικό γιατί αφορά και τις διεθνείς ε, υποχρεώσεις που έχουμε αναλάβει. Ορισμένες αρχίζουν να ισχύουν ε, από του χρόνου. Επίσης η αναθεώρηση των ευρωπαϊκών ε, εποπτικών αρχών. Και επίσης οι πανευρωπαϊκές ε, προσωπικές συντάξεις ε, που θα βοηθήσουν πολύ την ε, πρόθεση των κεφαλαίων αγορών και της Ένωσης Κεφαλαίων Αγορών και το ίντις για παράδειγμα δεν πρέπει να το ξεχάσουμε το συζητάμε τόσα χρόνια μήπως υπάρχει κάποια δυνατότητα συμφωνίας και ανέφερα διάφορα θέματα που αφορούν την Ένωση Κεφαλαίων Αγορών όλα αυτά θα βοηθήσουν οπωσδήποτε την ανάπτυξη, θα βοηθήσουν τις κεφαλαιαγορές, θα βοηθήσουν τη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας και άρα την οικονομική ανάπτυξη. Το θέμα είναι λοιπόν να αξιοποιήσουμε κατά το μέγιστον αυτές τις ευκαιρίες. Και τώρα νέες πρωτοβουλίες, βιώσιμη χρηματοδότηση, fintech. Και εδώ έχουμε τονίσει ότι η Ευρώπη θέλει να ηγείται της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής. Το είπαμε και στη Συμφωνία των Παρισίων. Άρα αυτή είναι η ευκαιρία να μετατρέψουμε τα λόγια μας σε πράξη, ιδιαίτερα στον τομέα και στον τομέα των ε, χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, επίσης για τις διαμεθοριακές συναλλαγές και συνεργασία. Να υπάρξει ενοποίηση του κλάδου που να βοηθήσει τους πελάτες. Και αυτή η πολύ καλή πρόταση. Να λοιπόν κάποιες προτεραιότητες αλλά δεν θέλω αυτό να εκλειφθεί ο ισχυρισμό ότι δεν είναι οι υπόλοιπε προτάσει σημαντικέ και δεν θα πρέπει να επιτύχουμε, να επιδιώξουμε να επιτύχουμε τη συμφωνία. Νομίζω ότι η προσέγγιση του Προέδρου, του Προέδρου Γκουαντιέρη είναι καλύτερη. Ας εργαστούμε με βάση αυτή την, ε, ε, ε, τη φιλοδοξία και θα δούμε τι θα επιτύχουμε. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ξέρω πως τα μέλη μας δουλεύουν σκληρά και είναι και πολύ αποτελεσματικοί, αλλά ναι. Σίγουρα και η σειρά προτεραιότητας που δώσατε καλύπτεται τα, καλύπτεται τα ίσως κάτι να λείψει, αλλά σίγουρα τα κόκκινα δάνεια και κάποια ακόμα θα ενταχθούν. Ξέρω ότι υπάρχει και ένα επίμαχο θέμα το οποίο πρόκειται να ανακοινώσετε, αλλά Άκουσα την ε, παρουσίασή σας και νομίζω ότι ε, τουλάχιστον ε, εκεί δεν θα υπάρξει πρόβλημα με το νομοθετικό πλαίσιο και με τις αμοιβαιοποιήσεις, αλλά ίσως αυτό που θα πρέπει να κρατήσουμε κατά νου είναι η ανάγκη του να είμαστε ρεαλιστές στις επιδιώξεις μας και καλό θα ήταν πριν καταθέσετε τις ίδιες προτάσεις να μας ζητήσετε να τις διαβάσουμε. Η κυρία Μπέρε, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Αντιπρόεδρε, πρέπει να σας πω πως αισθάνομαι έκπληξη. Καθένας από εμά θεωρεί πως ο δικός του φάκελος αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα γιατί τρέχει ο χρόνος. Και με κατέπληξε η απάντησή σας ε, στον κύριο Μπάλτς που είναι συντονιστής του ΕΛΚ και συνεισηγητής για την αναθεώρηση των οίκων εποπτεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί τον οίκων αξιολόγησης με γιατί δεν αναφερθήκατε στο θέμα αυτό. Νομίζω λοιπόν ότι έχετε 20 φακέλους ε, στο τραπέζι και δεν τους αναφέρατε. Γιατί? Γιατί αν εσείς δεν ε, ξεκινήσετε να επενδύετε σημαντικούς πόρους στο θέμα αυτό, δεν θα καταφέρουμε να το διεκπαιρεώσουμε. Και γνωρίζετε σε ποιο βαθμό για το μέλλον της Τραπεζικής Ένωσης και της αγοράς κεφαλαίων, το θέμα αυτό είναι σημαντικό. Και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι μπλοκαρισμένο στην ε, εισαγωγή σας. Ε, δεν το αναφέρατε, δεν το αναφέρατε και στην απάντηση στο συνάδελφό μου. Επίσης, πρόσφατα στείλατε μία ε, επιστολή ε, για τα διδάγματα και τις πληροφορίες που λάβατε από τα όσα συνέβησαν με την τράπεζα ABLV και για το γεγονός πως δεν έχετε ε, εργαλεία παρακολούθησης των συστημικών κινδύνων που ελοχεύουν στις τράπεζες λόγω του προβλήματος του ξεπλήματος χρήματος. Και την επόμενη μέρα που ξέσπασε η υπόθεση αυτή η Ντανιέλ Νούι η οποία είναι ε, υπεύθυνη για την εποπτεία των τραπεζών, μας είπε και σας είπε πως χρειάζεται να ε, του άρθρου 32 ε, και ε, ζητήσει της EBRD ε, και ζήτησε να γίνει. Αυτό δεν το αναφέρατε εσείς. Γιατί λοιπόν δεν αναφερθήκατε στο σημείο αυτό και τι στόχο έχετε μέχρι το τέλος της θητείας για να καλύψετε και αυτό το θέμα. Να ξεκινήσω με την πρώτη ερώτηση για την απάντηση που έδωσα στον κύριο Μπάλτς και στην ερώτησή του για τις προτεραιότητες. Είπα τις πρώτες τρεις προτεραιότητες και πιο συγκεκριμένα είπα το πακέτο για τις τράπεζες, τα εποπτικά και τα ΠΕΠ. Αυτή ήταν η πρώτη μου απάντηση προς τον κύριο Μπάλτς και νομίζω ότι αυτό έχει καταγραφεί και από τη γραμματεία της ΕΚΟΝ γιατί έχει καταγράψει τις απαντήσεις που σας έδωσα. Οπότε προφανώς ο εποπτικός ε, μηχανισμός θα αναθεωρηθεί ως ε, προτεραιότητα και ή και υποπτίας παράλληλα. Μην ανησυχείτε λοιπόν, θα σεβαστούμε το χρονοδιάγραμμα έτσι ώστε να πετύχουμε μια συμφωνία του χρόνου. Ε, και πάντα πριν λήξει η τρέχουσα θητεία. Το επαναλαμβάνω εδώ. Οπότε ναι. Μην ανησυχείτε, είναι προτεραιότητα το θέμα. Για τα εργαλεία που θα χρειαστούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο κατά του ξεπλήματος χρήματος, πρέπει να σας πω ότι είχαμε αρκετές υποθέσεις ε, στα κράτη-μέλη, την υπόθεση που αναφέρατε και αλλά και κάποιες άλλες που αποδεικνύουν ότι πρέπει να κινηθούμε. Και εμείς εργαζόμαστε για να βρούμε τρόπους να επιβάλλουμε την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ε, και πώς αυτό μπορεί να γίνει σε ε, όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε ε, και τα εργαλεία που δίνει η οδηγία και τα σχετικά με το ξέπλυμα χρήματος μπορούμε αυτά να τα επιβάλλουμε μέσω των σχετικών αρμοδίων αρχών και καλέσαμε την ΕΚΤ, το μηχανισμό και τις εποπτικές αρχές να ξεκινήσουν κοινέ προσπάθειες για να αντιμετωπίσουν αυτό το θέμα. Και με τον κύριο Τίμερμαντς και ε, την Επίτροπο Γιούροβα προετοιμάσαμε μια επιστολή ε, προς τον Μηχανισμό Εποπτείας, προς την ΕΚΤ, ε, καλώντας τους να ξεκινήσουν με το θέμα αυτό και ελπίζω πως εν ευθέτω χρόνο θα μπορέσω να σας παρουσιάσω πιο συγκεκριμένες ιδέες και προτάσεις. Οπότε θα πρέπει και την EBRD ε, στα πλαίσια του άρθρου 32. Έτσι δεν είναι. Ναι. Αυτή η αναθεώρηση είναι ένα σημείο που θα αξιολογήσουμε με την ΕΚΤ. Προκύπτει το θέμα της εναρμόνισης, ε, το θέμα της εκαθάρισης ε, τραπεζών που είναι σε πτώχευση. Οπότε αυτό είναι μόνο ένα από τα ζητήματα που θα συζητηθούν εκεί. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ καλά λοιπόν. Θα δούμε στην αξιολόγηση άλλων διατάξεων προβράσης της ΕΚΤ πάνω σε αυτό το άρθρο αν θα υπάρχουν κάποιες συνέπειες. Μπερτ Λούκεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα κύριε Επίτροπε. Μία από τις νομοθετικές πρωτοβουλίες που αναφέρατε για να βοηθήσουμε την ε, ανάπτυξη που, ε, που επιδιώκεται είναι πώς θα ρυθμίσουμε τις εταιρείες επενδύσεων που θέλει η Κομισιόν να φύγει από το CRR-CRD αν δεν έχουν συστημική σημασία και γι' αυτό θέλει να επιβάλλει λιγότερες ρυθμιστικές υποχρεώσεις αυτές τις επενδυτικές εταιρείες. Έχω όμως τώρα μία ερώτηση για την αντιμετώπιση των ε, μέσου μεγέθους ε, εταιρεών επενδύσεων όπου οι κεφαλιακές απαιτήσεις καθορίζονται με βάση τους λεγόμενους παράγοντες ΚΑΠΑ. Υπάρχουν ε, δύο δυνατότητες. Είτε θα καθοριστεί έτσι ο παράγοντας ΚΑΠΑ ούτω ώστε για τις εταιρείε αυτές οι κεφαλαιακές απαιτήσει να ανταποκρίνονται στις κεφαλαικές ε, απαιτήσει που επιβάλλονται στις τράπεζες που επίσης χειρίζονται τέτοια αξιόγραφα. Ή δεύτερον, η στάθμιση αυτού του παράγοντα ΚΑΠΑ θα καθοριστεί με βάση τις ανάγκες χρηματοοικονομικής σταθερότητας. Η, η EBA προτείνει την πρώτη προσέγγιση και η Κομισιόν ακολουθεί. Δηλαδή, η Κομισιόν ζητάει σχετικά υψηλέ κεφαλαιακές απαιτήσει για αμέσου μεγέθου εταιρείε επενδύσεων. Και από ό,τι φαίνεται, θέλει να υπάρξει ε, ισότητα συνθηκών ανταγωνισμού μεταξύ αυτών των εταιριών και των τραπεζών. Και δεν, δεν βασίζεται σε μία ανάλυση των κινδύνων για την ε, σταθερότητα των ε, και το ερώτημά μου, γιατί το έκανε αυτό η Κομισιόν, πιο συγκεκριμένα. Για ποιο λόγο, ποια είναι η δική αιτιολόγηση για να επιβάλλουμε σε αυτές τις εταιρείε επενδύσεων υψηλότερες κεφαλικές απαιτήσει από αυτές που θα επέβαλε η ανάγκη για σταθερότητα των αγορών. Δηλαδή, ποια είναι η ιεράρχηση των πολιτικών στόχων που κάνετε, ούτω ώστε να προστατεύονται οι τράπεζες έναντι αυτών των εταιριών που απλώς χειρίζονται αξιόγραφα. Καλώς όσον αφορά αυτό, αυτή την ερώτηση για τις επενδυτικές εταιρείες και την αναθεώρηση του τομέα πράγματι προτείναμε αναθωρημένο προληπτικό πλαίσιο για τις επενδυτικές επιχειρήσεις με στόχο να εξασφαλίσουμε αναλογική προσέγγιση και απαιτήσει κατά περίπτωση που για τα διάφορα επιχειρηματικά πρότυπα και τους ανάλογους κινδύνους. Πράγματι, κάναμε διάκριση μεταξύ συστημικά σημαντικών επενδυτικών εταιριών που παραμένουν εντός του πλαισίου του CRR-CRD, CRRD, κατηγορίας 2 ή κατηγορίας 3 είναι αυτές οι επενδυτικές επιχειρήσεις με συγκεκριμένο καθεστώς που, είναι διαφορετικά από το CRCD λαμβάνοντας υπόψη ε, μικρότερου βεληνικούς δραστηριότητες εξασφαλίζοντας επαρκή κάλυψη των κινδύνων και διευκολύνοντας και την είσοδο στην αγορά ταυτόχρονα και ανταγωνισμό σύμφωνα με τις απαιτήσει της ενώσεως των κεφαλαγορών. Οι απαιτήσει για μικρότερες εταιρείε θα είναι απλούστερες από ό,τι για μεγαλύτερες. Όσον αφορά τις πολύ μεγαλύτερες συστημικές επενδυτικές επιχειρήσεις, μέχρι τώρα δεν έχουμε κάποια στοιχεία που να δείχνουν ότι μη συστημικές επενδυτικές ε, εταιρείε μπορεί να καταλήξουν σε υψηλότερε απαιτήσει, μπορούμε να το συζητήσουμε, αλλά δεν έχουμε κάποια στοιχεία που να καταδεικνύουν κάτι τέτοιο. Εν πάση περιπτώσει, η πρότασή μας εμπεριέχει σταδιακή εφαρμογή των νέων διατάξεων για μη συστημικές επιχειρήσεις για να μειωθεί μεγάλη αύξηση των απαιτήσεων και φροντίζοντας να καλύπτονται και ακραίες περιπτώσεις εάν κάτι τέτοιο συμβεί σίγουρα εφαρμόζουμε την αρχή της αναλογικότητας και εδώ στην αναθεώρηση του τομέα των επενδυτικών εταιριών. Ευχαριστώ. Λιβ Βέρνικ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Επίτροπε, δέκα χρόνια πέρασαν από την τελευταία οικονομική και χρηματοστική κρίση και διερωτάται κανείς πότε θα έρθει η επόμενη κρίση. Δεν μπορούμε να το προβλέψουμε αυτό. Πρέπει αυτή τη, στιγμή, αυτή τη φορά να είμαστε προετοιμασμένοι. Η, η έκθεση την Παγκόσμια Οικονομική Σταθερότητα του Διεθνούς Ταμείου που δημοσιεύτηκε τον προηγούμενο μήνα ενετόπισε αυξανόμενους κινδύνους βραχυπρόθεσμους και μεσοπρόθεσμους. Τρεις ανησυχίες υπάρχουν. Πρώτα απ' όλα, ο συγχρονισμός σε παγκόσμιο επίπεδο ε, της τιμολόγησης που εκθέτει τα οικονομικά κέντρα και προθυμένε οικονομίες σε παγκόσμιες οικονομικές συνθήκε. συνθήκες. Δεύτερον, σε ένα περιβάλλον που αυξάνονται τα επιτόκια, ο κίνδυνο, της αύξηση τιμή των χρεογράφων ε, οφείλεται στη διακύμανση των, ε, της ρευστότητας ε, διαφόρες ποσοστά μόχλευσης. Και μετά έχουμε και την κυκλική φύση ε, της κατανομής των πιστώσεων που δημιουργεί κινδύνους ε, υπάρχουν αυτές οι ανησυχίες και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εν τη αυτή περιπτώσει πώς μπορούμε ε, να προστατεύσουμε το χρηματοπιστωτικό μας ε, σύστημα από ενδεχόμενους κλειδονισμούς από αυτά τα φαινόμενα. Απάντηση πράγματι. Είναι κάτι που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το τονίζει ότι τώρα η οικονομική περίοδος είναι καλή Έχουμε ανάπτυξη οικονομική για έκτο έτος και τα 28 κράτη-μέλη είναι σε οικονομική ανάπτυξη, έχουν επιστρέψει, η απασχόληση είναι σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, ε, η ανεργία είναι σε επίπεδα που υπήρχαν πριν την κρίση. Έχουμε θετικές εξελίξεις στην οικονομία, αλλά βλέπουμε ότι υπάρχουν και νέφοι στον ορίζοντα. Ε, δεν μπορούμε να περιμένουμε η οικονομική ανάπτυξη αυτή να συνεχιστεί επαόριστον ε, και γι' αυτό πρέπει να ενισχύσουμε την αντοχή των οικονομιών μας τώρα και του χρηματοστικού τομέα μας τώρα, τόσο ώστε να είμαστε σίγουρα προετοιμασμένοι για την επόμενη ε, κρίση όταν αυτή συμβεί. Επίσης, παρακολουθούμε τους κινδύνους αυτούς ε, που αναφέρατε για τον συγχρονισμό όσον αφορά την τιμή των κατοικιών, τις τιμές των αξιογράφων στην αγοροπολισία αυτών και άλλα στοιχεία. Δεν το κάνει αυτό μόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου. Κάποιους από τους κινδύνους αυτούς βλέπουμε ότι επηρεάζουν λιγότερο την Ευρωπαϊκή Ένωση από ότι άλλες προθυμένες οικονομίες, κατά μέσο όρο, ε, λιγότερες υπερτιμημένες τιμές των αξιογράφων δεν μπορούμε να αποκλείσουμε όμως ε, ενδεχόμενους ε, προβλήματα λόγω κινδύνων και αύξηση των τιμών των αξιογράφων. Ε, πρέπει να προετοιμαστούμε γι' αυτό. Εν γέννη, ο χρηματοπιστωτικό μας τομέας είναι πιο καλά προετοιμασμένος τώρα από ό,τι κατά παρελθόν για να αντιμετωπίσει αυτού του είδους τα προβλήματα. Έχουμε μεγαλύτερο απόθωμα απόσβεσης των κλειδονισμών στο χρηματοπιστωτικό τομέα σε περίπτωση μεγαλύτερων ποσοστών ρευστότητας κεφαλαίων, μικρότερη μόχλευση και ακόμα προσπαθούμε να ολοκληρώσουμε το ρυθμιστικό και το εποπτικό πλαίσιο. Γι' αυτό αναφέρθηκα στη σημασία του πακέτου αυτού για τις τράπεζες. Ε, και είναι σημαντικό στοιχείο που πρέπει να ολοκληρωθεί. Συνοψίζοντας, ε, πράγματι παρακολουθούμε αυτούς τους κινδύνους και συμφωνούμε με την εξολόγηση, Τώρα πρέπει να δραστηριοποιηθούμε για να εξασφαλίσουμε ότι η οικονομία μας και ο οικονομικός και χρηματοπιστωτικός τομέας μας είναι αρκετά ανθεκτικοί για να αντιμετωπίσουν αυτές τις ενδεχόμενες ε, προκλήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Παπαδημούλης. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, I will speak in Greek. Ε, σας ευχαριστώ για την ενημέρωση που μας δώσατε αλλά επιτρέψτε μου να σας ρωτήσω για τη χώρα μου, την Ελλάδα, καθώς πλησιάζουμε στην ολοκλήρωση του τρίτου και τελευταίου προγράμματος. Βρισκόμαστε στα τελευταία μέτρα για την ολοκλήρωση αυτής της δύσκολης πορείας και αυτή την ώρα έχει σημασία να εφαρμοστεί το Pacta Sunt Servanta από όλες τις πλευρές. Υπάρχει μια συμφωνημένη πορεία, ένας οδικός χάρτης που κατά το Eurogroup πρέπει να ολοκληρωθεί στις 21 Ιουνίου. Ολοκλήρωση της τέταρτης και τελευταίας αξιολόγησης με τα μνημονιακή στρατηγική, ελάφρυνση του χρέους, όπως έχει ήδη αποφασιστεί ως πλαίσιο από το Eurogroup τον Μάιο του 16 και τον Ιούνιο του 2017 και προσδιορισμός της μεταμνημονιακής εποπτείας με βάση τον κανονισμό 472. Επειδή κάθε καθυστέρηση στην υλοποίηση αυτού του συμφωνημένου πακέτου είναι επιζήμια γιατί ο χρόνος είναι χρήμα και προσθέτει η καθυστέρηση αβεβαιότητα, θα ήθελα να σας ρωτήσω δύο πράγματα. Το πρώτο, πριν από λίγες μέρες είπατε ότι οι αποφάσεις για την ελάφρυση του χρέους στη συμφωνημένη που δεν θα επιβαρύνουν ούτε ένα ευρώ τους Ευρωπαίους φορολογουμένους αλλά θα βοηθήσουν την Ελλάδα να ανακάμψει και να επιστρέψει στις αγορές είναι ζήτημα λίγων μηνών. Ορισμένοι στην πατρίδα μου στην Ελλάδα, που τους αποκαλώ Κασάνδρες, ισχυρίστηκαν ότι με τη δήλωσή σας εισηγήστε την αναβολή των αποφάσεων για μετά το Eurogroup της 21ης Ιουνίου. Θα ήθελα να μου, να μου διευκρινίσετε αυτή τη δήλωσή σας. Η Κομισιόν θέλει και εργάζεται για αποφάσεις της 21 Ιουνίου και για το χρέος. Και το δεύτερο, πώς σκοπεύει η Κομισιόν να συμβάλλει ώστε οι διαφορές μεταξύ Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και Ευρωπαίων Δανειστών να μην οδηγήσουν σε αναβολές και καθυστερήσεις σε βάρος της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας. Σας ευχαριστώ. Κύριε Παπαδημούλη, πραγματικά υπερβήκατε το πλαίσιο. Λοιπόν, ναι, αυτό αφορά άλλο τμήμα των αρμοδιοτήτων μου. Αλλά όντως είμαστε σε μια κρίσιμη περίοδο. Ολοκληρώνεται το ελληνικό πρόγραμμα Και σε γενικές γραμμές το πρόγραμμα ε, τα πάει καλά. Η Ελλάδα υπερεύει τους φορολογικούς της στόχους και μάλιστα με ουσιώδη τρόπο. Όπως διαπιστώσαμε για άλλη μια φορά πέρυσι. Και έχει αρχίσει η αξιολόγηση, η αποστολή είναι ήδη στην Αθήνα και ε, οι διαπραγματεύσεις γίνονται αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Συνολικά θα έλεγα ότι υπάρχει σαφής δέσμευση από όλες τις πλευρές από τους θεσμούς, από τις ελληνικές αρχές, να καταλήξει επιτυχώς το ελληνικό πρόγραμμα. Συζητάμε ε, κάποιες εκκρεμούσες ε, πρώτερες δράσεις και ορισμένα άλλα στοιχεία και κάποια θέματα που πρέπει να συζητήσουμε είναι και μέτρα για το χρέος. Και όπως είπα και δημοσίως πριν από μερικές μέρες, αυτή η εργασία, και το είπα δημοσίως, αυτή η εργασία συνεχίζεται και όταν ε, μίλησα για τους επόμενους μερικούς μήνες εννοούσα τον Μάιο και τον Ιούνιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται για να, διευκολύνει, να διευκολυνθεί αυτή η συμφωνία, να τηρήσει το χρονοδιάγραμμά της και πιστεύουμε ότι είναι εφικτό με βάση τις παραμέτρους που καθόρισε το Eurogroup, τους οποίους και εσείς αναφέρατε. Δεν θα υπάρξει δηλαδή ονομαστική, ονομαστικό κούρεμα, αλλά οι συνθήκες εξυπηρέτησης του χρέους θα αλλάξουν ούτως ώστε η Ελλάδα να επιτρέψει στις χρηματαγορές και να σταθεί στα πόδια της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν είναι πλήρως δεσμευμένη να υπάρξει αυτή η συμφωνία η οποία πρέπει να επιτευχθεί πριν από τη λήξη του προγράμματος. Τώρα για πώς εργαζόμαστε και πώς συνεργαζόμαστε με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Συνεργαζόμαστε επικοδομητικά, γιατί έχει συμμετάσχει μέχρι τώρα στο πρόγραμμα. Όχι μέσω απευθείας ε, συμμετοχής, οικονομικής συμμετοχής, αλλά με βάση κάποια, κάποιες προληπτικές ε, ρυθμίσεις. Συζητάμε λοιπόν για το τι μορφή συνεργασίας ή δέσμευσης θα, μπορούμε, θα μπορέσουμε να επιτύχουμε σε αυτή την τελική φάση του προγράμματος. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Βάλη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να κάνω δύο ερωτήσει στον Επίτροπο Ντομπρόσκης. Η πρώτη για το γνωστοτικό αυτό το πακέτο και κυρίως είμαι ικανοποιημένο διότι στην έκθεση Σίμονς η τονιστηκε αναγκαιοτητα να εγγυηθούμε support impact στις μικροσές επιχειρήσεις, να τις υποστηρίξουμε και για τον τομέα τον πράσινο και τον παράγοντα για την, κοινωνική, για την υποστήριξη. Να δώσουμε λοιπόν κάποιο περιθώριο όσον αφορά τι κεφαλοχικέ απαιτήσει. Για, την έκθεση Λούντ που ψηφίσαμε για την Τραπεζική Ένωση στο Κοινοβούλιο υπάρχει ένα τμήμα όπω και σε άλλε εκθέσει κατά το παρελθόν για την Τραπεζική Ένωση στο Κοινοβούλιο, που τονίζει και υπογραμμίζει τα χρεόγραφα του δευτέρου και τρίτου επίπεδου εντό των Ευρωπαϊκών Τραπεζών. Θα ήταν σκόπιμο να γίνει κάτι προ αυτή την κατεύθυνση, διότι πρόκειται περί αγοράς μεταξύ ε, το ύψος 7 δις ε, ευρώ όταν το σύνολο των, ε, κόκκινων δανείων είναι στα 900 με 910 δις. Θα ήθελα να ξέρω αν έχει πρόθεση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει κάτι ή μαζί με την Κεντρική Τράπεζα και τις μυστικούς φορείς να κάνει κάτι. Αναφερθήκατε επίσης στα ευρωμόλογα που που μάλλον συγγνώμη, τα ψεύτικα Eurobond που δεν ε, επιτρέπουν μερισμό των κινδυνών μεταξύ των χωρών. Θα ήθελα να ξέρω μήπως υπάρχει ένας κίνδυνος με μια τέτοια πρόταση τόσο στήρα όσον αφορά τον μερισμό των κινδύνων, μήπως υπάρχει ένα πρόβλημα μεγαλύτερο που θα αντιμετωπίσουμε στο μέλλον εν ώψη κλειδονισμών για την Ευρωζώνη. Διότι αν δεν έχουμε εργαλεία που μπορούν να διαχειριστούν την πίεση των αγορών θα πρέπει να χειριστούμε μια κρίση πάλι με μεταρρυθμίσεις πάρα πολύ λίγο, πάρα πολύ δημοφιλής με μειώση των αμοιβών. Είναι θεμελιώδης όπως ε, ε, είπε και ο Ντράγκη στη Φλωρεντία στην τελευταία του ομιλία να βρούμε μια λύση για τον επιμερισμό των χρεών και των βαρών. Διαφορετικά κάποιες χώρες σε επόμενη κρίση θα μπορούσαν να καταστραφούν και ε, ε, ή να θέλουν να απομακρυνθούν. Χρειάζονται μεταρρυθμίσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση για να δούμε αν πρέπει να ακολουθήσουμε προς μια κατεύθυνση ή τελικά οι λαοί τελικά θα κινηθούν στη θέση μας. Θα ήθελα να εξετάσουμε το ενδεχόμενο μιας διεξόδου ε, όσον αφορά τα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσει το σύστημα της Ευρωζώνης. Σας ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις αυτές και για την πρώτη να σας πω πως μάλλον πρόκειται για σχόλιο περισσότερο για το παράγοντο αυτά της κοινωνικής στήριξης. Ξέρετε πως εμείς αυτή την πρωτοβουλία την στηρίζουμε και συνεργαζόμαστε με τον εισηγητή κύριο Σίμων για να βρούμε κάποιες πιο συγκεκριμένες λύσεις. Αυτή τη στιγμή σχεδιάζουμε αυτή τη στήριξη, την πράσινη στήριξη ε, η οποία θα είναι παρόμοια με τη στήριξη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δηλαδή ε, οριακές μειώσεις κεφαλαϊκές απαιτήσει όταν οι τράπεζες δανείζουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πρέπει όμως να διατηρήσουμε κατά νου υπάρχει ε, και την προληπτική διάσταση όταν λέμε πράσινη δεν θεωρείται ε, ότι είναι και ακίνδυνη μια επένδυση οπότε ε, κάπου πρέπει να διατηρήσουμε και μια απόσταση ασφαλείας. Τώρα για τις ερωτήσεις που κάνατε που ήταν πολλές για τη δράση επίπεδου 3 που είναι κομμάτι της εποπτικής ε, ε, δράσης για την μείωση του κινδύνου σε αυτά τα ε, στοιχεία ενεργητικού να σας πω πως την ανακοίνωση για την Τραπεζική Ένωση από πέρσι τον Οκτώβριο έχουμε δώσει κάποια στοιχεία Νομίζω ε, έχετε στο μυαλό σας το βιβλίο επενδύσεων των χαρτοφυλακίου, με συγχωρείτε, των τραπεζών που πολλές φορές συμπεριλαμβάνονται ε, κάποιοι κίνδυνοι. Να σας πω πως αυτό αποτελεί κομμάτι ε, του τραπεζικού πακέτου ήδη από το 2016. Ε, επίσης, γίνονται κάποιες ε, συζητήσεις για τη στάθμιση αυτής της απαραίτητης αναθεώρησης στα πλαίσια της Συμφωνίας Βασιλεία οπότε θα δούμε ποια είναι η σωστότερη προσέγγιση, πάντως θα αποτελέσει κομμάτι των προτασιών μας. Τώρα για τα... Ε, για τις ομολογίες, ε, τα κρατικά ομόλογα ε, που ε, στηρίζονται από αξιόγραφα και από τίτλους, να σας πω πως αυτή είναι μία λύση ε, την οποία θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε για να λύσουμε κάποια κενά που υπάρχουν στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών γιατί τους έχουμε ζητήσει να κάνουν μια διαφοροποίηση ε, στα επενδυτικά τους ε, χαρτοφυλάκια και να μην επενδύουν μόνο ε, στις δικές τους ε, αγορές κρατικών ομολόγων. Οπότε εδώ θα μπορούσαμε να έχουμε ένα ε, διαφορετικό προϊόν που θα βασίζεται σε κρατικές ομολογίες από όλα τα 19 κράτη-μέλη. Ξέρω πως ε, όλοι αντιμετωπίζουν την πρόταση αυτή με ιδιαίτερη φυλακτικότητα. Υπάρχουν ε, και κρατημέλη και εμπλεκόμενοι ε, που ε, ανησυχούν γιατί θεωρούν πως μπορεί να αποτελέσει ε, ένα πρώτο βήμα για αλλαγή στην αντιμετώπιση ε, αυτών των χαρτοφυλακίων για πρόταση η οποία προσπαθεί να επιφέρει μια και καλυμμένη εναρμόνιση αλλά όχι δεν σημαίνει κάτι τέτοιο και έχουμε ζητήσει να γίνει μια αξιολόγηση της πρότασης αυτής βασιζόμενη μόνο στα ιδιαίτερα της στοιχεία. Ο κύριος Μονό. Ευχαριστώ. Στα πλαίσια του Παγκόσμιου Εμπορικού Πολέμου, ε, όποια και να είναι η Αμερικανική διοίκηση, είτε είναι δημοκράτες είτε ρεπουμπλικάνοι, μας δημιουργούν στρατηγικά προβλήματα σε επίπεδο ε, ευρωπαϊκών ε, επιχειρήσεων. 9 δις 9 πρόστιμο στην BNP, Γαλλική Τράπεζα, γιατί η Αμερικάνη έδωσε μια ε, ερμηνεία πραγματική, πραγματικά περίεργη για το τι σημαίνει ε, πρόστιμο. Γιατί όχι στην Κούβα και στο Ιράκ και στην BNP ε, Παριμπά. Τώρα, για την Λετονική Τράπεζα ε, να σας πω ότι ε, χρεοκόπησε γιατί είπαν οι Αμερικάνοι ότι σκέφτονται ε, ενδεχομένως να επιβάλλουν πρόστιμα στην ABLV. Ε, και τι έγινε στην περίπτωση αυτή. Μίλησε η κυρία Μπερές για το θέμα του υποπτικού μηχανισμού και τα προβλήματα που είχαμε εδώ. Και είχαμε και αυθαίρετες ε, κυρώσεις εναντίον της Ρουσάλ, μια ρώσικης επιχείρηση παραγωγής αλουμινίου για παράδειγμα, που μπορεί αυτό να οδηγήσει σε αδυναμία αποπληρωμής των χρεών της επιχείρησης αυτής στις διεθνείς αγορές που μπορεί να μας φέρει σε μία ε, αντίστοιχη ε, ε, κρίση στην αγορά με αυτή που είχαμε το 2008. Τώρα, κυρώσεις στο Ιράν. Και πάλι αυθαίρετες κυρώσεις που θα τιμωρήσουν τις δικές μας εταιρείε λόγω της αυθαίρετης απόφασης μια ξένης δικαιοδοσίας. Τώρα, η Άλστρομ. Θυμόσαστε τι έγινε όταν έπεσαν έξω η Enron και η WorldCom το 2003, λέει ο μιλητής. Τι θα γίνει αν μια μεγάλη ε, ε, ενεργειακή ή ε, ευρωπαϊκή εταιρεία ή μια αυτοβιομηχανία ε, ευρωπαϊκή πέσει έξω το 2018 γιατί έβαλαν κάποια πρόστιπα οι Αμερικάνοι. Φανταστείτε τι έγινε με την ABLV και φανταστείτε τι θα γίνει αν μια εταιρεία ευρωπαϊκή δεν μπορεί να κεφαλοποιηθεί παρόλο που κυρώσει ακόμα δεν έχουν επιβληθεί. Αυτό σημαίνει ότι ε, θα αποσταθεροποιηθεί απολύτως η ε, ευρωζώνη με τις ε, συνέπειες που μπορούμε όλοι να φανταστούμε. Αυτό το EU Blocking Regulation θεωρώ ότι είναι ένα αγγελικό κείμενο που δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τους συστηματικούς, συστημικούς κινδύνους που αντιμετωπίζουμε. Και είδατε τι κάνουν οι Αμερικάνοι στην Ευρώπη. Εσείς αυτό το συστημικό κίνδυνο τον παίρνετε ε, ε, σοβαρά υπόψη. Ο πρόεδρος ε, της σχετικής επιτροπής ε, της ΕΚΤ ανησυχεί. Οπότε θέλω να μου πείτε πώς μπορείτε εσείς να βοηθήσετε σε αυτό το επίπεδο την Ευρώπη που κινδυνεύει. Λοιπόν, πολύ περίπλοκη ερώτηση που μου θέσατε. Υπήρξαν κάποιες δυσχέρειες στις εμπορικές μας σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο μονομερών ε, κυρώσεων σε προϊόντα χάλιβος και αλουμινίου μετά την 1η Ιουνίου. Ξέρετε ότι πήραμε κάποιες παρατάσεις ε, καθυστέρηση της επιβολής αυτών των κυρώσεων ως Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θέλουμε μια μόνιμη λύση. Δεν είναι δυνατόν από μήνα σε μήνα να αποφασίζονται αυτές οι περαιτέρω εξαιρέσει από την επιβολή κυρώσεων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και άλλοι ευρωπαϊκοί θεσμοί λοιπόν είναι σε πολύ στενή επαφή με τους συνομιλητές μας από τις ΗΠΑ για να αντιμετωπιστεί αυτή η ανησυχία. Τώρα, κατόπιν, αναφερθήκατε στο Ιράν. και την ε, καταγγελία της συμφωνίας με το Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την αποχώρησή τους από αυτή τη συμφωνία. Αυτό μας ανησυχεί ως Ένωση. Είναι επικίνδυνο προηγούμενο. Κάποιες χώρες μονομερώς ε, να αποχωρούν από διεθνείς συμφωνίες. Παρά το ότι η... ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας επανειλημμένα έχει βεβαιώσει ότι το Ιράν συνεχίζει να τηρεί τη συμφωνία και έχει περιορίσει το πυρηνικό του πρόγραμμα στο βαθμό που απαιτεί Και αξιολογούμε αυτή τη στιγμή τις οικονομικές επιπτώσεις και τα άλλα ενδεχόμενα αποτελέσματα των Αμερικανικών κυρώσεων κατά του Ιράν και τις εξωεδαφικές τους επιπτώσεις σε ενωσιακές εταιρείε και ιδιαίτερα στον χρηματοπιστωτικό μας τομέα και επιχειρήσεις αυτού του κλάδου. Όπως είπατε, ο κανονισμός EU blocking έχει περιορισμένη επίπτωση σε αυτή την περίπτωση λόγω του διεθνούς χαρακτήρα του τραπεζικού συστήματος και της έκθεσης ιδιαίτερα των μεγάλων συστημικών τραπεζών στο αμερικανικό οικονομικό σύστημα και των συναλλαγών του σε δολάρια. Δύσκολα θέματα. Αυτά πρέπει λοιπόν να αντιμετωπιστούν και εξετάζουμε αυτή τη στιγμή τον τρόπο με τον οποίο θα το αντιμετωπίσουμε. Τώρα, αυτά που είπατε για την εφαρμογή των κανόνων κατά του ξεπλήματος χρήματος, τονίζω ότι πρέπει να έχουμε αξιόπιστη και συντονισμένη πολιτική για το ξέπλυμα χρήματος σε ενωσιακό επίπεδο για να εντοπίσουμε αποτελεσματικά αυτές τις ανησυχίες εντός της Ένωσης χωρίς να περιμένουμε δράσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Ευχαριστώ πολύ. Ryan Hayes. Κύριε Αντιπρόεδρε, σας ξανακαλωσορίζω στην Οίκον. Η Επιτροπή δημοσίευσε ένα πρόγραμμα για το πρόγραμμα δράσης για τις ε, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες για τους καταναλωτές. Έχουμε ενιαία αγορά για τις εταιρείε του κλάδου, αλλά όχι για τους καταναλωτές. Οι διαμεθοριακές ε, δραστηριότητες για ενυπόθηκα δάνεια, ασφαλής κτλ. είναι πολύ χαμηλό. Ποιε ε, δραστηριότητες θα προωθήσετε κατά προτεραιότητα μέχρι το τέλος της θητείας για να υπάρξει περισσότερη πρόοδος, περισσότερη φιλοδοξία. Στη χώρα μου έχουμε μέσο επιτόκιο 3,2 ενώ στην Ένωση είναι ένα και κάτι κατά μέσο όρο. Πρέπει να σταματήσουν να υπάρχουν αυτοί οι φραγμοί για το καθεστώς αξιολόγηση, για το καθεστώς φερεγγιότητας. Με αυτόν τον τρόπο θα μειώσουμε το κόστος, θα μειώσουμε τις τιμές για να πάρουν οι καταναλωτές μας ό,τι χρειάζεται με τον καλύτερο τρόπο. Ποιε δραστηριότητες, ποιε προτεραιότητες θα έχετε σε αυτό το τομέα. Το πρόγραμμα δράση δηλαδή των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών για του καταναλωτέ. Και δεύτερον, ξέρετε πόση δουλειά έγινε από το κοινοβουλίο μα για να επιτευχθούν συμβιβασμοί για την ε, μεταρρύθμιση των χρηματαγορών. Υπάρχει λοιπόν τώρα κανονισμό, λειτουργεί, σημαντικό κανονισμό, όλοι τον δεχόμεθα και θα είναι σημαντικό για να μειωθούν οι συστημικοί κίνδυνοι. Αλλά υπολοιπόμεθα των ΗΠΑ, άρα είναι σημαντικό να επιτύχουμε σωστή ρύθμιση. Αλλά ξέρετε ότι κάποιοι συνάδελφοι σα έγραψαν ότι η ΕΣΜΑ ε, ε, απαγόρευσε το λεγόμενο share conciliation και reverse actions. Όμω, δεν υπάρχουν προτάσει τη ευρωπαϊκή επιτροπή γι' αυτό. Καμία τροποποίηση. Και ξαφνικά στην ΕΣΜΑ βλέπουμε μια υποσημείωση, συμφωνεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτή η πρακτική απαγορεύεται. Σημαντική λοιπόν ερώτηση. Είναι λογικό να ληφθεί απόφαση επίπεδου 1 στο επίπεδο 2 οι συνομοθέτες, δηλαδή αυτοί που εκλέγονται για να παίρνουν τις αποφάσεις, αγνοούνται. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Ε, okay. So on the first uh, question... Για την πρώτη ερώτηση για τις σηματοστικές υπηρεσίες ε, των καταναλωτών και το σχετικό σχέδιο δράσεως. Ανέφερα μια συγκεκριμένη πρόταση νομοθετικού περιεχομένου για διασυνοριακές πληρωμές που επεκτείνει την αρχή αυτή των ευρωπαϊκών πληρωμών σε εσωτερικές, σε χώριες τιμές σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελπίζουμε λοιπόν και η Επιτροπή Οικονομική να ασχοληθεί με το θέμα και να εξασφαλίσει την έγκριση ε, της πρότασης μέχρι τέλος της θητείας. Θα έχει απτά ωφέλη για τους καταναλωτές ε, από αυτή την ε, ολοκλήρωση σε αυτό το τομέα. Πέρσι το Δεκέμβριο συστάθηκε ομάδα εργασίας. Ομάδα εμπειρογνωμόνων. Θέμα της. Οι υποχρεώσεις για τον πελάτη. Ε, από μακριά ε, ψηφιακή ταυτοποίηση και άλλες δυνατότητες. Ένα από τα εμπόδια για τη συνοριακή παροχή χρηματοστικών υπηρεσιών είναι η γνώση για τον πελάτη. Να γνωρίζει κανείς τον πελάτη. Και θέλουμε να το διευκολύνουμε αυτό να συμμορφωθούν οι τράπεζες με αυτή την απέτηση γνώσης του πελάτη και σε διασυνοριακό επίπεδο. Σε αρκετού τομεί έχουμε προτάσεις. Προτάσεις για την άρση των διασυνοριακών εμποδίων για την παροχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Αναφέρθηκα στο PEPS για τα προσωπικά προϊόντα συντάξεων που είναι πολύ ανεπτυγμένα σε κάποιες χώρες και πολύ λιγότερα ανεπτυγμένα προϊόντα αλλού και αν, έχουμε, αν περάσει η πρότασή μας για πανευρωπαϊκά συνταξιδοτικά ε, πακέτα, είναι, αυτό είναι υποφελές για τους καταναλωτές. Είναι περισσότερο, ε, δεν ανήκει τόσο στον τομέα της ε, Λιανικής, αλλά της Κεφαλογικής Ένωσης, της Ένωσης των Κεφαλογορών. Αλλά είναι σημαντικό για τους καταναλωτές. Από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι θα δοθεί μια φιλόδοξη συνέχεια στο σχέδιο δράσης για τις σηματοστικές υπηρεσίες για τους ε, ιδιώτες. Τώρα, για τις χρηματαγορέ και, και κοινή, το μηχανισμό της κοινή δήλωσης. Έγιναν κάποιες συζητήσεις και υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κυρίως η Νομική Επιτροπή, έκανε ανάλυση και επιβεβαιώνει την άποψη που εξεφράστη από τις ε, προπτικούς φορείς ότι μηχανισμός για την ε, εξίες και τις ε, μετοχές δεν συνάδει με τον κανονισμό, με τον πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και η νομική υπηρεσία αποφάσισε να γνωμοδοτήσει σχετικά με το θέμα αυτών των μετοχών να δημοσιοποιήσει σύμφωνα με, τις, ε, με το πλαίσιο για την ε, διαβίβαση πληροφοριών προς τους πολίτες. Οπότε συνεχίζονται οι προσπάθειες μαζί με τους εμπλεκόμενους ε, φορείς. Σας ευχαριστώ. Έχουμε συζητήσει και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τις διαφορετικές απόψεις όλων για το θέμα. Και νομίζω ότι αυτό επιβεβαίωσε και η δική μας νομική υπηρεσία. Ο κύριος Φερνάντες παρακαλώ. Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι μεγάλη χαρά που σας έχουμε εδώ κύριε Αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Νομίζω ότι είναι σημαντικό αυτές τις συγκρίσεις να τις χρησιμοποιήσουμε όχι μόνο για να ε, παρακολουθούμε τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά για να κάνουμε και μία δημόσια παρακολούθηση ε, των θεμάτων αυτών για να γνωρίζουν και να ενημερώνονται οι εκλογείς μας για τα όσα συμβαίνουν εδώ. Ο κανονισμός που παρουσιάσατε εσείς στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο πριν από δυόμιση χρόνια πια έφτασε την ηλικία των 30 μηνών είναι το ίμιση της θητείας και πρέπει να σου πω ότι είναι σε κατάσταση αδιεξόδου ε, απόλυτης παραλυσίας και εδώ και στο Συμβούλιο με πέντε μήνες όπου δεν έχουμε κάνει καμία συνεδρίαση των σκιωδών γιατί τελευταία, την τελευταία φορά που συναντήθηκαν οι σκιώδεις μιλάω για το έντες εντάξει ήταν η 13η Δεκεμβρίου του περασμένου έτους πέντε μήνες και δεν έχουμε καμία ημερομηνία ε, στα χαρτιά μας για να συνεδριάσουμε μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Οπότε, επειδή κάνουμε αυτή τη σύγκριση, ήθελα να πω στους πολίτες που μας παρακολουθούν. Κάποιοι που είμαστε εδώ αισθανόμαστε ντροπή που εμείς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορούμε καν να προχωρήσουμε στις συζητήσεις αυτές ενός φακέλου του Ίντες που είναι πάρα πολύ σημαντικός. Γιατί Έχουμε το κοινό ψήφισμα, έχουμε την κοινή εποπτεία, τραπεζική ένωση, έχουμε το κοινό ρυθμιστικό πλαίσιο για τις τραπεζικές οντότητες, αλλά αν κάποια τράπεζα έχει πρόβλημα λόγω της τραπεζικής εποπτείας της Ευρώπης, ποιος θα πληρώσει, ο καταθέτης του κράτους μέλους ή ο προϋπολογισμός του κράτους μέλους, μόνος. Και δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Οι ευρωπαϊκές αρχές αποφάσισαν να εκαθαρίσουν τον Banco Popular και αν δεν είχε βρεθεί αγοραστής, οι Ισπανοί καταθέτες θα είχαν πληρώσει για μια απόφαση την οποία πήραν οι Βρυξέλλες. Και οι Πορτογάλοι θα είχαν πληρώσει. Έχει αυτό νόημα. Ή θα προχωρήσουμε ή ας πάμε εκεί που ήμασταν παλιά. Κάποιοι κατάφεραν να συζητήσουν μεταξύ τους και να προτείνουν διαφορετικές συμπληρωματικές πρωτοβουλίες, πρώτα απ' όλα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να συνεχίσουν οι διαπραγματεύσεις. Το ξέρετε κύριε Επίτροπε ε, η Γκουε εμείς προσπαθήσαμε να διαπραγματευτούμε με τους φιλελεύθερους, με το ΕΛΚ, με όλους, το Δεκέμβριο. Και μέχρι σήμερα δεν έχουμε λάβει καμία απάντηση. Και το χειρότερο είναι πως το Συμβούλιο πρόκειται να συνεδριάσει τον επόμενο μήνα, να δούμε αν συμφωνήσουν σε πολιτικό επίπεδο και θα φτάσει καθυστερημένα στο ραντεβού το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και χωρίς να έχει κάνει τη δουλειά τους. Και τι θα πούμε εμείς του πολίτες για τους οποίους είμαστε εμείς εδώ και οι οποίοι πληρώνουν την παρουσία μας εδώ. Uh, well, uh, on this um, uh, I can only agree, of course, from... Να συμφωνήσω βέβαια και εγώ εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Λυπάμαι πραγματικά που έχουμε τόσο περιορισμένη πρόοδο από το 2015 στο φάκελο Ίντις. Και ξέρετε κι εσείς πως είχαμε αξιολογήσει ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους ε, καθυστερεί αυτή η πρόταση. Και ποια είναι τα, ποιοι είναι οι ηθικοί κίνδυνοι που προκύπτουν. Ξέρετε πως πέρσι τον Οκτώβριο προτείναμε και εμείς κάποιες νέες ιδέες και κάναμε και μια συνάντηση για να συζητηθούν. Να δούμε πώς μπορούμε το ίντις να ενσωματωθεί, να ξεκινήσει πιο σταδιακά ας πούμε με την πρώτη φάση να στηρίζει τη ρευστότητα χωρίς όμως την κλοποίηση ζημίας και μετά υπό οι προϋποθέσεις για να περάσουμε από το στάδιο 1 στο στάδιο 2 το οποίο θα σήμαινε αυξημένη, ε, αυξημένο σύστημα ευρωπαϊκής τιτλοποίησης και από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής η φιλοδοξία μας είναι να μιλήσουμε, να μιλήσουμε για ένα σύστημα ευρωπαϊκό πλήρες αλλά αν θέλετε μπορούμε εμείς να σας διευκολύνουμε έτσι ώστε να δούμε ποια είναι τα ενδεδειγμένα βήματα έτσι ώστε να κινηθούμε προς αυτό το στόχο. Εν πάση περιπτώσει ελπίζουμε πως οι δικές μας ιδέες τις οποίες καταθέσαμε πέρυσι μπορεί, μπορούν να σας βοηθήσουν και να αποτελέσουν τη βάση για έναν ενδεχόμενο συμβιβασμό. Στο Συμβούλιο αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι γίνονται ε, οι τεχνικές εργασίες και πρέπει να πω πως προχωράνε αρκετά καλά. Έγινε μια συναδρίαση της ad hoc ομάδας εργασίας και έχουμε τη δική μας ανακοίνωση για τη συμπλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης η οποία εκκίνησε νέες συζητήσεις. Οπότε η Βουλγαρική Προεδρία εργάζεται ε, πάνω σε τεχνικά σημεία που έχουν να κάνουν με την πρώτη φάση. Σε πολιτικό επίπεδο δε, απόψεις των κρατών μελών αποκλίνουν μεταξύ τους. Όμως εμείς ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή είμαστε ακόμα δεσμευμένοι υπέρ αυτής της πρότασης και θα θέλαμε να σας βοηθήσουμε να επιτύχετε ένα συμβιβασμό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Πρέπει να σας πω κι εγώ ότι μου είναι πολύ δύσκολο να δικαιολογήσω όχι το γεγονό ότι υπάρχουν διαφορετικέ απόψει, αυτό είναι φυσιολογικό, αλλά το γεγονό ότι δεν κάνουμε συνεδριάσει για να συζητήσουμε αυτέ τι απόψει. Αυτό είναι απαράδεκτο. Μπορεί κάποιος να διαφωνήσει, αλλά ο δικός μας στόχος εδώ είναι να εργαστούμε έτσι ώστε να βρίσκουμε κάθε φορά ένα συμβιβασμό, όποιος και να είναι αυτός ο συμβιβασμός. Μετά ψηφίζονται, εγκρίνονται, δεν εγκρίνονται, αλλά αυτή η ε, παραλυσία δεν είναι σωστή. Και είναι και άδικη. Ο κύριος Κίρτσος, παρακαλώ. Thank you, Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Αντιπρόεδρε, Μπορείτε να συνοψίσετε για μας ποιες είναι οι εξελίξεις ε, με το Brexit στο χρηματοστοπιστικό κλάδο. Μας είπατε πως εκεί κινείστε γρήγορα. Έχετε να μας δώσετε πληροφορίες σχετικά με τα θέματα τα οποία αντιμετωπίσατε και τα θέματα τα οποία ακόμα ε, είναι προς επίλυση. Και έχω και μια δεύτερη ερώτηση για τη μείωση του κινδύνου και τον επιμερισμό του κινδύνου που αποτελεί και τη βάση της Τραπεζικής Ένωσης. Λόγω των γεγονότων στην Ιταλία, ο κίνδυνος έχει αυξηθεί και νομίζω ότι έτσι του ερμηνεύουν και οι αγορές γιατί τα επιτόκια αργά αλλά σταθερά αυξάνονται για την Ιταλία, για την Ελλάδα επίσης και βέβαια πολλά κράτη δεν επιθυμούν να κάνουν επιμερισμό του κινδύνου, ούτε η Γερμανία, ούτε η Αυστρία, ούτε οι κατοχώρες. Οπότε πώς θα καταφέρετε να συμφιλιώσετε αυτές τις εξελίξεις που κατά τη γνώμη μου δεν είναι και πολλά υποσχόμενες. Okay. Ε, so, ε, Κοιτάξτε, όσον αφορά το πρώτο ερώτημά σας για το Brexit, συνεχίζονται οι διάφορες διεργασίες. Θα επικεντρωθούμε και επί του χρηματοστοτικού τομέα που είναι η δική μου αρμοδιότητα σχετικά με αυτό. Τι κάναμε λοιπόν τους προηγούμενους μήνες. Δημοσιεύσαμε ανακοινώσεις προετοιμασίες όπως αποκαλούνται, περιγράφοντας αναγκαίες προετοιμασίες που πρέπει να εφαρμοστούν από διάφορους συμμετέχοντες στην αγορά, από θεσμικούς φορείς, πώς θα προετοιμαστούν για τα διάφορα ενδεχόμενα σχετικά με το Brexit. Και υπάρχει συμφωνία για την δημιουργία μιας ομάδας υπό την ηγεσία της Τραπέζης της Αγγλίας και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας εξετάζει ενδεχόμενους κινδύνους και διάφορα ενδεχόμενα που άπτονται του Brexit. Ε, για τις 30 Μαρτίου του 2019 την ημερομηνία του Brexit συμπεριλαμβάνοντας επίσης τις διάφορες συνέπειες ε, σε περίπτωση μη συμφωνίας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ομάδα μας η διαπραγματευτική θέλει να, να γίνει μια τακτική ε, έξοδος της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει πολιτική συμφωνία περί μεταβατικής περίοδου που θα βοηθήσει να διασκεδαστούν κάποιες ε, ανησυχίες και να ανακουφιστούν κάποιες χρονικές πιέσεις, αλλά η μεταβατική αυτή περίοδος, εν πάση περιπτώσει, αποτελεί τμήμα της συμφωνίας απόσυρσης. Χρειάζεται συμφωνία στα, πάνω σε αυτό στα πλαίσια της συμφωνίας απόσυσης του Ηνωμένου Βασιλείου. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις όπως και το θέμα των Ιρλανδικών συνόρων και πώς αντιμετωπιστεί αυτό και αυτό συνδέεται στενά και με τις μελλοντικές τελειωνιακές μας σχέσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο. Οπότε συνεχίζονται οι διαργασίες. Είναι σημαντικό να σημειωθεί πρόοδος διότι ο Μάρτιος του 2009 είναι πρώτον πυλών. Σε λιγότερο από ένα χρόνο θα φτάσει αυτή η ημερομηνία. Η άλλη ερώτηση ίσως για τη μείωση του κινδύνου, τον επιμερισμό των κινδύνων, για τις εξελίξεις στα κράτη-μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Ιταλίας. Όπως γνωρίζετε δεν σχολιάζουμε ε, τις διαδικασίες ε, σχηματισμού κυβερνήσεων ή πολιτικά θέματα στα κάτι μελη Ασχολούνται τα κάτι μελη με αυτά σύμφωνα με τις συνταγματικές τους διαδικασίες. Αυτό που τονίζουμε όμως είναι ότι είναι σημαντικό να υπάρχει δημοσιονομική πειθαρχία και κυρίως στην περίπτωση της Ιταλίας να μειωθεί το δημοσιονομικό έλλειμμα και το δημόσιο χρέος. Αυτά είναι σημαντικά στοιχεία. Είναι παράγοντες κινδύνου που επηρεάζουν την οικονομία. Συζητήσαμε το θέμα με την παρούσα Ιταλική κυβέρνηση, συμφωνήσαμε όσον αφορά την δημοσιονομική πορεία για το τρέχον έτος και αυτό είναι και το μήνυμα που απευθύνουμε προς τη νέα κυβέρνηση ότι είναι σημαντικό να παραμείνει σε αυτή την πορεία και η νέα κυβέρνηση. Ευχαριστώ. Πολ Τάγκ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε που είσαστε εδώ. Η Επιτροπή Οικονομική υιοθέτησε την έκθεση πρωτοβουλίας για τη βιώσιμη, ε, ε, τα βιώσιμα χρηματοπιστωτικά. Θα σας στηρίξει το Κοινοβούλιο στις προσπάθειές σας, το Ευρωκοινοβούλιο εκφράστηκαν ανησυχίε και ευχέ. Θέλουμε να αλλάξει ο χρηματοστικό τομέα και δεν ξεκίνησαν καν οι αλλαγέ. Ερώτηση. Η αλλαγή που προτείνεται πότε, Μάιο 23 Μαΐου, 24 Μαΐου, οι αλλαγές που προτείνεται καλύπτουν ένα αρκετά ευρύ πεδίο. Να δώσω κάποια παραδείγματα γιατί ανησυχούμε. Για, πρα για τα, για τα πράσινα στοιχεία ενεργητικού και την ταξινόμηση αυτών. Δεν συμπεριλαμβάνονται άλλοι παράγοντε που είναι σημαντικοί. Το ESG, Φερρυπίν. Η παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, παραβίαση δικαιωμάτων εργαζομένων, φορολογικό σχεδιασμό. Αν ξεκινήσετε με τα πράσινα στοιχεία ενεργητικού, τι θα κάνετε με του άλλου παράγοντε που τονίζει το, το Κοινοβούλιο. Δεύτερον, δεν συμπεριλαμβάνεται η ιδέα των την πρόταση του ESRB για ε, μια ε, προληπτική πολιτική που λαμβάνει υπόψη και το κλίμα. Κεφαλουχικές απαιτήσει, επίπεδα εκθέσεις λαμβάνονται υπόψη. Ε, αυτά λαμβάνονται υπόψη. Μετά, τρίτον, και θα πρέπει οι επενδυτές να λαμβάνουν υπόψη όχι μόνο τις οικονομικές συνέπειες των κινδύνων, αλλά και τους κινδύνους που, ε, που δημιουργούνται για εκείνους τους οποίους εκπροσωπούν. Ε, γιατί αυτός ο κίνδυνος των γιατί με συμπλαμβάνονται και οι τράπεζες που είναι πολύ σημαντικές όσον αφορά τον οικονομικό τομέα. Έτσι έχουν τα πράγματα. Γιατί να μην γίνει ευρύτερη κάλυψη, όπως είναι οι χειριστές των στοιχείων ενεργητικού, τα συντεξιωτικά ταμεία, και όσα σχετίζονται γενικά με τις τράπεζες. Ευχαριστώ για τη στήριξή σας. Για το πρόγραμμα δράσης για βιώσιμη χρηματοδότηση. Θέλουμε να έχουμε φιλόδοξους και ευρύς στόχους και παρακολούθηση της ε, επίτευξής τους. Έχουμε εκπονήσει μια έκθεση που θα αποτελέσει τη βάση για την συνέχιση εξέτασης της εφαρμογής των βασικών συστάσεων του προγράμματος δράσης για να καλύψουμε όσο πιο ευρύ φάσμα τομέων γίνεται. Τώρα, για το πώς θα, ταξινομήσουμε τα διάφορα στοιχεία προτείνουμε να υπάρξει μια δομή διακυβέρνησης για την ταξινόμηση, την ιεράρχηση. Όταν θα δημιουργηθεί, θα γίνει κατόπιν η συγκεκριμένη ταξινόμηση. Και τονίζουμε ότι η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής θα πρέπει να είναι ο πρώτος μας στόχος από πλευράς αυτής της ιεράρχησης είναι κρίσιμη σημασία για να προωθήσουμε την πράσινη πλευρά της βιώσιμης χρηματοδότησης. Αλλά κατόπιν θα επεκταθούμε και σε άλλους τομείς. Και θέματα περιβαλλοντικής, κοινωνικής και, διακυβέρνη... και πλευράς διακυβέρνησης, ESG. Αυτή λοιπόν η δομή διακυβέρνηση, όπω λέμε, θα αντιμετωπίσει πρώτα τα θέματα κλιματική αλλαγή, αλλά κατόπιν θα διευρύνει το πεδίο δράση τη. και σε άλλους τομείς. Για τα στοιχεία ενεργητικού τα οποία έχουν παραμεληθεί, θέλουμε να μειωθούν ε, οι κίνδυνοι για τέτοια στοιχεία ενεργητικού. Θα δούμε τι παρακάτω, παραπάνω μπορούμε να κάνουμε για τις ε, καταπιστε, καταπιστευματικές ανάγκες ε, και τις υποχρεώσεις των ε, επικεφαλής ε, και άλλων υπευθύνων για τις περιουσίες ατόμων που επενδύουν και που κάνουν διάφορες επιλογές. Δεν είναι αυτές οι, οι δραστηριότητες ε, οι πιο συνήθεις των τραπεζών. Για τους συνήθεις πελάτες, αν έχεις απλώς ένα λογαριασμό ταμιευτηρίου και έναν τρέχοντα, δεν σου προσφέρουν και πολλές δυνατότητες ε, επενδύσεων σε διάφορα χρηματοπιστωτικά προϊόντα. Αν όμως η τράπεζα αρχίζει να σου δίνει και ατομικές συμβουλές, ούτως ώστε να είναι ιδιωτική τραπεζική, ιδιωτικές τραπεζικές συμβουλές, αυτές που δίδονται σε κάποιους πελάτες, τότε πρέπει να διευκρινίσουμε και να καθορίσουμε τι υπηρεσίες μπορούν να παρέχουν οι τράπεζες. Στοχεύουμε λοιπόν να έχουμε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα παρακολούθησης τις δράση μας σε στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ούτως ώστε όλα αυτά τα θέματα να αποτελέσουν αντικείμενο συμφωνίας και να εφαρμοστούν κατά την τρέχουσα θητεία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ ο Τόμας Μα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Αντιπρόεδρε, ακούσατε ότι στηρίζουμε ιδιαίτερα πολύ ημών πολλές από τις ιδέες. Να, εδώ κάθομαι. Εδώ. Και είπαμε σαφώς και τι μπορεί να επιτύχει και το ίδιο το Κοινοβούλιο. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικές οι εκθέσεις που προωθούμε. Τι γίνεται με την περαιτέρω εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει να υπάρχει ένα πλαίσιο προστασίας των καταθετών σε ευρωπαϊκό επίπεδο αν ε, χρεοκοπήσει μια τράπεζα. Αλλά δεν θέλουμε ε, οι ζημίες να γίνονται κοινέ για όλους. Δεν είναι δυνατόν να λέγεται κάτι τέτοιο εύκολα. Ξέρετε ότι άκουσα ότι το συνολικό ποσό που θα μπορούσε να αφορούν αυτά τα μέτρα είναι 760 δις. Τι πρόκειται να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και όχι απλώς να πει ότι κοιτάξτε πολλά πρέπει να τα κάνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ποιος ε, θα εγγυηθεί ότι στο τέλος οι καταθέσεις των αποταμιευτών και το χρήμα των φορολογουμένων δεν θα αντιμετωπιστούν με λάθος τρόπο για να σωθούν κάποιες τράπεζες. Στην Ιταλία ξέρουμε τι γίνεται τώρα με, την, το σχηματισμό της κυβέρνησης. Τι μπορούμε να κάνουμε. Οι δεξιοί λαϊκιστές θέλουν να κάνουν κυβέρνηση. Είναι ιδιαίτερα ε, λυπηρό αυτό. Και ακούσαμε ε, ότι η πρώτη τους απέτηση είναι ότι θέλουμε μια ελάφρυνση 230 δισεκατομμυρίων. Δεν ξέρω τι θα πούνε οι Έλληνε γι' αυτό. Βλέπω ότι τα ελληνικά ομόλογα, συγγνώμη, τα ιταλικά ομόλογα πιέζονται. Η πιστοληπτική ε, ικανότητα των ιδρυμάτων γίνεται όλο και πιο επισφαλής και η Κεντρική Τράπεζα συνεχίζει να αγοράζει αλίπητα ιταλικά ομόλογα. Κάνατε ό,τι μπορείτε δεν είναι τμήμα της ε, Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στα πλαίσια της ε, ανεξαρτησίας της να ε, λάβει τις σωστές αποφάσεις και να το πει. Βεβαίως θέλουμε να μειωθεί το χρέος κάθε χώρας, αλλά δεν είναι δυνατόν να πούμε ότι θα τους το χαρίσουμε. Αυτό δεν το κάναμε σε άλλες χώρες. Δεν μπορεί να γίνει και στην περίπτωση της Ιταλίας. Λοιπόν, Ε, να απαντήσω λοιπόν για την ε, ερώτηση του έτης και της απώλειας ε, τιτλοποίησης, όπως επίσης της μείωσης των κόκκινων δανείων στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών. Και αν υπάρχει κάποιος πιο σταδιακός τρόπος να εισάγουμε την ίδις, ξεκινώντας με μία ε, στήριξη της ρευστότητας και μετά με μία δεύτερη φάση με την, ε, ε, με την τίτλοποίηση και την στήριξη των κόκκινων δανείων. Να σας πω πως για τα κόκκινα δάνεια, τα στοιχεία που έχουμε, οδηγούν στο 910 δις ευρώ στα χέρια ευρωπαϊκών τραπεζών. Βέβαια υπάρχουν και διαφορετικές μεθοδολογίες υπολογισμού από τις διάφορες πηγές. Εν πάση περιπτώσει έχουμε μια σημαντική μείωση ε, της αναλογίας από το 6,7% των κόκκινων δανείων που ήταν ε, στην ακμή της κρίσης στο Ζενίδη στο 4,4% σήμερα, αλλά τα ενημερωμένα στοιχεία θα τα έχουμε διαθέσιμα αύριο. Οπότε ίσως τα στοιχεία που σας δίνω σήμερα δεν είναι τα πιο πρόσφατα και αύριο ενδεχομένως θα δούμε κάτι πιο ενημερωμένο. Μετά, για τα 230 δις αλληλευθρύνσης ε, χρέους που ετήθηκε ε, από τα κόμματα τα οποία πρόκειται να σχημητήσουν κυβέρνηση γιατί είχαμε μια διαρροή ε, πάνω στην οποία βασίζεται αυτός ο αριθμός και έχει να κάνει με ένα παλιό σχέδιο κειμένου που δεν ισχύει πια Οπότε νομίζω ότι αυτό δεν αποτελεί κομμάτι ε, του προγράμματος ε, σχηματισμού κυβέρνησης στη χώρα. Και θα ήταν και παράδοξο αυτό γιατί ε, είναι στοιχεία ενεργητικού της ιταλικής ε, κρατικής συγχωρείτε, της ε, Ιταλικής Κεντρικής Τράπεζας που βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, οπότε θα ήταν παράδοξο να ζητήσουν κάτι τέτοιο. Αλλά ξέρετε, πολλά από αυτά τα οποία διαβάζουμε είναι παράδοξα. Όπως επίσης ε, η μείωση του φόρου του συντελεστή που θα επιβάλλεται στους πιο πλούσιους κατοίκους. Ξερδική ιδέα, τι να πω. Η κυρία Γκίλ, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Κύριε Αντιπρόεδρε, χαιρετίζω τη δέσμευσή σας ώστε να έχουμε βιώσιμη, ε, ένα βιώσιμο χρηματοπιστωτικό κλάδο και με χαρά θα διαβάσω και τις προτάσεις σας την επόμενη εβδομάδα και για την ταξινόμηση, την κατηγοριοποίηση. Νομίζω ότι πρέπει να είναι φιλόδοξα τα σχέδιά σας ε, και σύμφωνα με την έκθεση Scott το ε, που υποβάλαμε εμείς. Τώρα για τους παράγοντες για τη διακυβέρνηση θα ήθελα να μου πείτε τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Τα, θα τα κάνετε σε αυτή τη θητεία, θα είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα, θα έχουμε ελάχιστους κοινωνικούς και κυβερνητικούς ε, κανόνες και κατόφλια, θα τα δούμε μεσοπρόθεσμα, μακροπρόθεσμα ή μόνο βραχυπρόθεσμα από σήμερα. Γιατί πρέπει να εξασφαλίσουμε πως η πράσινη χρηματοδότηση θα αποτελέσει τον κανόνα και όχι ε, ε, το ελάχιστο σε σχέση με το 99,9% της μη βιώσιμης χρηματοδότησης που υπάρχει σήμερα. Και τι θα κάνετε. Και περνώ στο δεύτερο σημείο. Χτες συζητήσαμε το σχέδιο έκθεσης για τους προληπτικούς κανόνες για τις επενδυτικές εταιρείε. Και ο συνομοθέτης εδώ στις διαπραγματεύσεις MIFID ήταν το πλαίσιο ισοδυναμίας να καλύπτει όσο το δυνατόν μεγαλύτερες επενδυτικές και χρηματοδοτικές δυνατότητες για όσους συμμετέχουν στην ευρωπαϊκή αγορά ε, κεφαλαίων. Κάποιοι θέλουν, να περιορίσουμε το πεδίο εφαρμογή τη ισοδυναμία έτσι ώστε να μειωθεί η δυνατότητα συμμετοχή κάποιου είδου επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στα πλαίσια λοιπόν του Brexit, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αξιολογήσει την επίπτωση αυτού του περιορισμού συμμετοχή και τι σημαίνει αυτό για την Ευρωπαϊκή Ένωση, μια και ε, το ίμιση αυτών των εταιριών βρίσκεται στο Ηνωμένο Βασίλειο σήμερα και ε, δίνει κάποιες εναλλακτικές δυνατότητες χρηματοδότησης που δεν υπάρχουν σε αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είπατε πως θα πρέπει ο ιδιωτικός κλάδος να εξασφαλίσει πως οι συμβάσεις θα συνεχίσουν να τρέχουν ομαλά χωρίς ε, αναταραχές. Μπορούν οι ίδιες οι αγορές να λύσουν αυτό το πρόβλημα. Τι σκοπό έχετε, πώς μπορεί να αντιμετωπίσει μόνο η αγορά όταν δεν υπάρχει ξεκάθαρο ρυθμιστικό πλαίσιο. Τι κάνετε, κάνατε, συναντηθήκατε με τον Υπουργό Οικονομικών, συναντήσατε την Κεντρική Τράπεζα τη Αγγλία και αν ναι, ποια ήταν τα αποτελέσματα αυτών. Και τέλος, για να επανέλθω απαντήσατε στον Brian Hayes και το καταλαβαίνω ε, για τις εταιρείες, τις αγορές ε, κεφαλαίων. Αν αυτό θεωρείται τόσο σημαντικό, γιατί δεν το εντάξατε καταρχήν στην πρόταση έτσι ώστε να συζητηθεί με τον κατάλληλο τρόπο. Uh, okay. Καλώς. Πράγματι, πολλές ερωτήσεις ετέθησαν. για βιώσιμο χρηματοδοτικό τομέα και ταξινόμηση όπως είπα για την αλλαγή του κλίματος και την επέκταση και σε άλλους παράγοντες ε, διακυβέρνησης και κοινωνικούς παράγοντες. Το θέμα είναι πότε. Εξαρτώνται όλα αυτά από το νομοθετικό έργο. θα κάνουμε νομοθετικού περιεχομένου πρόταση, αλλά δεν θα συμπεριλάβουμε την ταξινόμηση αυτή καθεαυτή, αλλά θέματα δομή διακυβέρνηση τη ταξινόμησης. Στο σχέδιο δράση ακολουθούμε, εάν πραγματοποιηθεί αυτό που θέλουμε που είναι αισιόδοξο, και αν το νομοθετικό έργο ολοκληρωθεί εντός ενός έτους, εάν γίνουν αυτά, θα έχουμε τιμή, ε, στο τρίτο τρίμηνο του 2019 έτοιμη την ταξινόμηση. Ίσως είναι λίγο αισιόδοξη αυτή η προοπτική που περιγράφω. Εξαρτάται από τις νομοθετικές διαδικασίες. Αν ακολουθήσουν το χρονοδιάγραμμα είναι εφικτό. Δεν μπορώ να προδικάσω τώρα επακριβώς την ταχύτητα πορείας των εργασιών για την ταξινόμηση. Πάντως αυτό είναι το σχέδιο, αυτή είναι η κεντρική ιδέα αντιμετώπισης του ζητήματος. Ήδη το συζητήσαμε και πριν αυτό. Θέλουμε να έχουμε ένα ευρύ σχέδιο δράσεως που θα καλύπτει διάφορους τομείς χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών εξασφαλίζοντας τη χορήγηση κινήτρων στον χρηματοπιστωτικό τομέα και συμπεριφορά να κινηθεί προς πρότυπα και στόχους ε, που λαμβάνουν υπόψη την πράσινη προσέγγιση του κλίμα. Τώρα την εξέταση των επενδυτικών εταιριών και το σχετικό πλαίσιο διακυβέρνησης από αυτού προέβημε σε αξιολόγηση αντιχτύπου. Κάναμε μια αξιολόγηση της πρότασής μας πρώτα απ' όλα δεν περιορίζουμε τους κανόνες περί ισοδυναμίας. Θέλουμε να δούμε ποια κριτήρια χρησιμοποιούνται για την απόφαση περί ισοδυναμίας. Είναι ευρύτερο το θέμα. Διερευνούμε την ισοδυναμία σαν ενδεχόμενο πλαίσιο χρηματοπιστωτικής συνεργασίας, οικονομικής συνεργασίας με το Ηνωμένο Βασίλειο. Μέχρι τώρα το ιστορικό της Ευρωπαϊκή Ενώσης όσον αφορά την ισοδυναμία είναι καλό πάνω από 200 αποφάσεις περί ισοδυναμίας που αφορούν 30 νομικά καθεστώτα των μεγαλύτερων οικονομιών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται περισσότερο από άλλη μεγάλη οικονομία, περισσότερο στι ισοδυναμίε της Ευρωπαϊκής Ένωση από ότι άλλε δικαιοδοσίε. Και η ισοδυναμία θα παίξει σημαντικό ρόλο, πιστεύω, και στις οικονομικέ μα σχέσει με το Ηνωμένο Βασίλειο. Η ιδέα δεν είναι να περιορίσουμε το καθεστώς των ισοδυναμιών, αλλά να καταλήξουμε σε σαφήλιση, συμπεφωνημένη για τις ισοδυναμίες. Και θα μπορέσουμε να, νομίζω πέρσι είχαμε ετοιμάσει ένα έγγραφο ή το 2016. Πέρσι, πέρσι. Εκεί περιγράφαμε την προσέγγισή μας όσον αφορά τις ισοδυναμίες την περίοδο μετά το Brexit. Το άλλο ερώτημα. Για την συνέχεια που θα δοθεί στις συμβάσεις. Εξαρτάται όσον αφορά τα παράγωγα και τις συμβάσεις περί ασφαλίσεων μπορούν να εφαρμοστούν διάφορες λύσεις από τον τομέα. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να βρεθούν λύσεις σε εθνικό επίπεδο μπορεί να βρεθούν λύσεις. Μπορεί να μεταφερθούν αυτές οι συμβάσεις σε φορείς εντός, που έχουν έδρα εντός Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Για τα παράγωγα και πρόσβαση σε διάφορα προϊόντα, κάποιοι κίνδυνοι αντιμετωπίζονται από το στα σταδίου 2. Και αν προσαρμοστεί δεόντως ο τομέας, μπορεί να βρεθεί μια προσέγγιση για άλλες υποδομές αγορές όπως ε, καταθετήρια παραγόγων εκεί το πρόβλημα μικρότερης κλίμακας και ο κίνδυνος για τη χρηματοπιστωτική ισορροπία και σταθερότητα μπορεί να αντιμετωπιστεί με άλλο τρόπο και σταδιακή εξάλληψη κάποιων μέτρων αν χρειαστεί. η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Τράπεζα της Αγγλίας και αρμόδιες ομάδες εργασίας αυτών μπορούν να επεξεργαστούν το θέμα αφορά τις συνέπειες απόσχησης, διαφοράς, χάσματος και θέλουμε να, να μην υπάρξει αυτό μετά το Brexit. Δεν ξέρω μετά τι να προσθέσω Δεν ξέρω τι απάντηση να δώσω για το θέμα των MFF. Συζητήθηκε από τους συνομοθέτες το θέμα, δηλαδή να επιτρέψουμε την ακύρωση επιμερισμού των κινδύνων σε αυτές τις συμφωνίες είναι κάτι που απορρίφθηκε από τους συνομοθέτες. Είναι ένα από τα επιχειρήματα που χρησιμοποιεί η νομική υπηρεσία περιγράφει την εικόνα λέγοντας ότι αυτή η πρακτική δεν ταιριάζει με τους ισχύοντες κανόνες και κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Η γνωμοδότηση και αξιολόγηση νομικής υπηρεσίας είναι δημοσία διαθέσιμη. Δεν ξέρω αν μπορώ να προσθέσουμε πολλά πράγματα πάνω σε αυτό σε αυτή τη φάση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για την παρουσία σας. Λοιπόν, να επανέλθω στο πρώτο θέμα που συζητήσαμε. Πόσο χρόνο έχουμε. Και αυτό μας περιορίζει τη δυνατότητα να περάσουμε πολλά νομοθετήματα. Αλλά δεν είναι μόνο θέμα χρόνου πολλές φορές το πρόβλημα. Αναφέρθηκε το έντις. Να μιλήσω γι' αυτό. το σύστημα εγγύησης ε, καταθέσεων. Δεν νομίζω πως το πρόβλημα είναι τεχνικές ε, διχογνωμίες ή διαφωνίες για το χρονοδιάγραμμα. Είναι θέμα εμπιστοσύνης μεταξύ κυβερνήσεων και εμπιστοσύνης ε, σε κάποια σημαντικά εργαλεία που έχουμε εφαρμόσει. SSM ή ακόμη και το CRD Άρα αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί. Το θέμα ότι δεν υπάρχει επαρκής εμπιστοσύνη. Οπότε, Ναι, υπάρχουν και άλλα θέματα που δεν είναι θέμα τεχνικών ε, διαφωνιών, αλλά έλλειψης εμπιστοσύνης. Και τι μπορείτε να κάνετε εσείς ως Επιτροπή όχι μόνο για να αντιμετωπίσετε τις τεχνικές δυσκολίες, αλλά για να επανέλθει η εμπιστοσύνη για τόσο σημαντικά θέμα, για παράδειγμα η αξιοπιστία του SSM, του CRD και διαφόρων άλλων. Απάντηση. Κοιτάξτε, πρέπει να επιτύχουμε την ισορροπία μεταξύ μείωσης κινδύνων και ενίσχυσης της εμπιστοσύνης, ούτως ώστε να υπάρξει επιμερισμός των κινδύνων. Νομίζω ότι οι Υπουργοί Οικονομικών συμφώνησαν το 2016 για το λεγόμενο οδικό χάρτη μείωσης κινδύνων. Τα περιέχει όλα αυτό το, αυτός ο δικός χάρτης για τη μείωση των κινδύνων. Και με βάση αυτό έχουμε υποβάλει τις προτάσεις μας για τους επόμενους στόχους. Όπως η πρόταση που κάνει το 2016 για το πακέτο για την Τραπεζική Ένωση. Έχει υπάρξει σημαντική πρόοδος για τη μείωση των κινδύνων, όπως περιγράφεται στον οδικό χάρτη που συμφώνησαν οι Υπουργοί Οικονομικών της Ένωσης. Πιστεύουμε λοιπόν ότι αυτή είναι η βάση για να σημειώσουμε τώρα πρόοδο και για τον επιμερισμό των κινδύνων. Βλέπουμε ότι οι συνθήκε είναι όριμες για να επιτευχθεί συμφωνία για μια τελική λύση, backstop, για ένα ενιαίο ταμείο εξυγένση και για το πρώτο στάδιο του έντις. Έχουν γίνει αυτές οι συζητήσει. Εδώ και χρόνια γίνονται. Τι σημαίνει μείωση κινδύνων, τι σημαίνει επιμερισμός κινδύνων. Πρέπει λοιπόν να τονίσουμε ότι ήδη έχουμε επιτύχει αρκετά ουσιώδη για τη μείωση των κινδύνων που μπορεί, μπορούν αυτά τα επιτεύγματά μας να προωθήσουν και, την περαιτέρω, και περαιτέρω την, ε, τον επιμερισμό των κινδύνων. Βέβαια, κοιτάξτε, υπάρχει θέμα εμπιστοσύνη, υπάρχει και θέμα προκαταλήψεων ορισμένε φορέ, λέει ο Πρόεδρο. Πολύ σημαντικό. γιατί κάπου διάβασα ότι αν είχαμε εφαρμόσει τα τελευταία χρόνια το έντις τότε κάποιες χώρες του Νότου θα ήταν καθαρή συνεισφορή στους προπολογισμού των, ε, της ε, Γερμανίας και της Ολλανδίας. Άρα υπάρχουν και προκαταλήψεις. Άλφρεντ Σάντα. Ευχαριστώ και καλημέρα. Πρώτη ερώτηση. Πρώτα απ' όλα, η ανάπτυξη των κρυπτονομισμάτων συζητιούνται στις Βρυξέλλες. Και εσείς τον περασμένο Φεβρουάριο συμμετείχατε σε μια συζήτηση στο Κυρίς Τραπέζι για τα κρυπτονομίσματα. Υπάρχει πολύ σκεπτικισμός για αυτά. Κυρίως ασχολούμεθα με τους κινδύνους από τη χρήση τους και όχι από τις ευκαιρίες. Αλλά κάποια συμβόλαια παραγών δεν είναι από πλευράς ε, των μικροεπενδυτών λιγότερο επικίνδυνα. Και ο τομέας των υπηρεσιών μπορεί να υποφεληθεί από τα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων. Άρα τι πλεονέσματα, πλεονεκτήματα θα προέκυπταν από τη χρήση αυτών των κρυπτονομισμάτων και πώς ε, αξιολογείται την εξέλιξη στα κράτη-μέλη για τα θέματα αυτά. Δεύτερη ερώτηση. Η πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ιδίω στον νότο τη Ευρώπη σε χρηματοδότηση ή βασίζεται στα παραδοσιακά τραπεζικά μοντέλα. Και οι εισαγωγέ στο χρηματιστήριο μικρομεσαίων είναι το ίμιση αυτών που γίνονταν πριν την κρίση. Πρέπει να κάνουμε λοιπόν περισσότερα για να υποστηρίξουμε την εισαγωγή του στι δημόσιε χρηματαγορέ. Πρόσφατα η Κομισιόν ξεκίνησε μία δημόσια διαβούλευση για το θέμα αυτό. Τι μέτρα προτίθεται να πάρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τι, αν είναι δυνατόν κάτι, θα μπορούσε να καταλήξει πριν το τέλος της θητείας. Και η τρίτη μου ερώτηση σχετίζεται με αυτό που είπε η κυρία Γκίλ για τους ασφαλιστές και τα συνταξιδοτικά ταμεία που έχουν συμβόλια στο Ηνωμένο Βασίλειο και αντίστροφα. Δηλαδή δικά μας που έχουν συμβόλαια στο Ηνωμένο Βασίλειο και αντίστροφα. Όπως ξέρετε αυτά τα συμβόλια εξαρτώνται από την άδεια που έχουν οι επιχειρήσεις να ε, έχουν συναλλαγές και στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπου και αν πάνε οι διαπραγματεύσει για τον Brexit, μπορείτε να πείτε στους πολίτες και του καταναλωτέ της Ένωσης που έχουν συμβόλαια με βρετανικές εταιρείε ότι θα μπορέσουν να αποφεληθούν από τα συμβόλαιά τους. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία λοιπόν. για τα κρυπτονομίσματα να ξεκινήσω με αυτά λέγοντας πως το θέμα αυτό το είδαμε και στο σχέδιο δράσης για τη FinTech. Δηλαδή πώς αντιμετωπίζουν τα νομίσματα αυτά οι ευρωπαϊκές αρχές και νομίζω ότι με τον τρόπο αυτό ε, έχουμε βάλει στα σκαριά καινούργιες εξελίξεις έτσι ώστε να αποφύγουμε αυτά τα κρυπτονομίσματα και να δούμε και ποια είναι τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν. Γνωρίζουμε πως υπάρχουν κάποιοι κίνδυνοι και οι ευρωπαϊκές ε, εποπτικές αρχές μετά από δικό μου αίτημα ε, προειδοποίησαν εκ νέου τους καταναλωτές για τους κινδύνους που κρύβουν, κρύβουν αυτά τα κρυπτονομίσματα, ε, για το ποιες είναι οι επενδύσεις και για το ότι δεν ε, υπάρχει καμία εγγύηση για αυτές τις επενδύσεις, έχει να κάνει καθαρά με προσφορά και ζήτηση και υπάρχει μεγάλη ε, πιθανότητα απώλειας ολόκληρης της ε, επένδυσης σε αυτά τα κρυπτονομίσματα. Πρέπει να σας πω πως και ο όρος ο ίδιος, κρυπτονόμισμα, ίσως να είναι παραπλανητικός. Γιατί η ΕΚΤ, για παράδειγμα, έχει τονίσει αρκετές φορές πως υπάρχει μόνο ένα νόμισμα στην περιοχή του ευρώ και είναι το ευρώ. Οπότε μπορείτε να το πείτε ε, κρυπτο κάρτες, κρυπτο επιταγές, κρυπτοβάουτσερ, αλλά δεν είναι κρυπτονόμισμα. Πάντως αυτά τα κρυπτο ε, στοιχεία ενεργητικού έχουν κάποια στοιχεία τα οποία ενδεχομένως θα αντιμετωπιστούν ε, νομοθετικά γιατί κάποια εμπίπτουν σε συγκεκριμένα νομοθετικά πλαίσια. Τώρα, μην ξεχνάτε πως υπάρχουν και διατάξεις για την καταπολέμηση του ε, ξεπλήματος βρώμικου χρήματος, οπότε όσοι παρέχουν ε, τέτοιου είδους κρυπτονομίσματα θα πρέπει να σέβονται τη σχετική νομοθεσία. Βλέπετε λοιπόν πως υπάρχουν αρκετές προεκτάσεις τις οποίες θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε όταν συζητάμε τις εξελίξεις με αυτά τα κρυπτονομίσματα. Τώρα για την ε, εισαγωγή των ε, μικρομεσαίων νομίζω ότι μέσα στο μήνα θα λάβετε τις σχετικές ε, προτάσεις και εμείς θα διευκολύνουμε τις μικρομεσαίες να μπουν στα χρηματιστήρια, να βγουν στις αγορές και θα χρησιμοποιήσουμε τους σχετικούς δείκτες με ευελιξία. Είναι μία από τις προτεραιότητές μας και βρίσκεται και στην ενδιάμεση ε, αναθεώρηση ε, ως στοιχείο και θα μπει και στην ε, πρόταση που θα καταθέσουμε σχετικά με τα θέματα της Νομισματικής Ένωσης τον Μάιο. Ένα από τα θέματα τα οποία σχολιάζουμε είναι αυτό των ε, συμβάσεων για τα παράγωγα και το συζητάμε σε επίπεδο εποπτικών αρχών επίσης. Συγγνώμη για την παράταση των συμβάσεων εν ώψη Brexit. Ε, εμείς εκεί έχουμε και μια ομάδα εργασίας που προσπαθεί να απαλύνει τις επιπτώσεις που θα έχει το Brexit, αλλά οι διαπραγματεύσεις ακόμα τρέχουν και υπάρχουν δύσκολα εκρεμή θέματα, οπότε σε αυτή τη φάση διστάζω από το να σας προσφέρω κάποιες εγγυήσεις γιατί επαναλαμβάνω οι διαπραγματεύσεις τρέχουν και τα αποτελέσματα δεν είναι ακόμα 100% σαφή. Βεβαίως προσπαθούμε να κινηθούμε προς μια ρυθμισμένη εξοδό η οποία θα ελαχιστοποιήσει ε, τις αναταραχές σας. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω πως ε, η συζήτηση όπως αναμένεται ήταν εξαιρετικά πλούσια. Μια πολύ θετική ανταλλαγή απόψεων. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ κύριε Επίτροπε, Επίτροπε Ντομπρόφσκης και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που ήρθατε. Η Επιτροπή μας τους τελευταίους αυτούς μήνες που μένουν θα δουλέψει σκληρά για να προσπαθήσει να κλείσει όσο δυνατόν περισσότερους φακίλους γίνεται και αν είναι δυνατόν όλους. Αυτός είναι ο στόχος μας και ελπίζω πως όλοι οι συνάδελφοι θα συνεργαστούν. Χρειάζεται να κάνουμε σκληρή δουλειά. για να βελτιώσουμε τη δυνατότητα να έχουμε ένα νομοθετικό πλαίσιο που θα προσφέρει και στον τομέα της ανάπτυξης αλλά και στην ε, σταθερότητα Συνάδελφε, συνάδελφε, τελείωσε ο χρόνος. Και πρέπει να συνεχίσουμε με το επόμενο σημείο της ημερής σας διάταξης. Η δική σας ε, πολιτική ομάδα είχε χρόνο να μιλήσει, όπως και όλες οι υπόλοιπες. Σας ευχαριστώ λοιπόν Επίτροπε και περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερής σας διάταξης.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 Yeah.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 So, dear colleagues, let's move to point 11. Αγαπητοί συνάδελφοι, το σημείο 11 της μέρας διάταξης. Να καλωσορίσω τον κύριο Ζαν Πολ που το γνωρίζετε όλοι πολύ καλά και τον εκτιμάτε. Είναι διακεκριμένος πρώην συνάδελφος. Τώρα μας επισκέπτεται ως πρόεδρος της ε, συμβουλευτικής ομάδας για την υποβολή χρηματοοικονομικών εκθέσεων. Είναι μαζί του και ο κύριος Άντριου Βότσμαν που είναι επικεφαλής εκτελεστικός και πρόεδρος της ε, ομάδας τεχνικών εμπειρογνωμών. Όπως ξέρετε τα λογιστικά θέματα τα τελευταία χρόνια παίζουν σημαντικό ρόλο στην εργασία της ΕΚΟΝ. Η δέσμευσή μας ε, στον τομέα το λογιστικό αντανακλάται με τη δημιουργία μια ομάδα εργασία. Την ομάδα, μόνιμη ομάδα για το IFRS που θέλει να συμμετέχει το Κοινοβούλιο όσο πιο νωρί γίνεται στην ε, εξέλιξη των διεθνών πιστοτικών προτύπων και την έγκρισή τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ΕΦΡΑΚ μαζί με το Ίδρυμα IFRS και το PIOB λαμβάνουν ε, συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριο αίτημα του Κοινοβουλίου για την παράταση της συμφωνίας για το Ίδρυμα ήταν να υπάρξει η δυνατότητα τακτικών ακροάσεων για να ενημερωνόμεθα για την εξέλιξη των ε, λογιστικών προτύπων. Οπότε ε, αυτή η ακρόαση είναι σε αυτά τα πλαίσια. Είναι ιδιαίτερα επίκαιρη γιατί το ΕΦΡΑΓ αυτή τη στιγμή διατυπώνει τις προτάσεις του για το νέο πρότυπο ασφαλίσεων IFRS 17 που ε, αναμένεται τον προσεχή Δεκέμβριο και το Κοινοβούλιο αναμένεται να εγκρίνει και ψήφισμα για το θέμα αυτό το οποίο θα παίξει ρόλο στη διαδικασία για τις συμβουλές για τον επιστογράφηση. Οπότε, αγαπητέ Ζαν Πολ, ε, σας δίνω τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Είμαι ευτυχής που είμαι εδώ. Είναι τιμή για μένα να, παρουσι... να είμαι παρίσταμε. Πρόεδρος τη Επιτροπής αυτής επί δεκαετία και βλέπω γνωστά πρόσωπα, φιλικά πρόσωπα. Σας ευχαριστώ αυτή την ευκαιρία που μας δίνει, μας δίδεται να έρθουμε να σας ενημερώσουμε από αυτού που κάνετε Φραγκ και τις διάφορες σκέψεις όσον αφορά τις προδιαγραφές που συζητούνται κυρίως τα FRS 17 Ανέλαβα τη δέσμευση όταν ήρθα για ακρόαση αυτή την επιτροπή το Μάιο του 2016 να ενισχυθούν οι σχέσεις με το Ευρωκοινοβούλιο. Προσπάθησα να το κάνω αυτό. Ελπίζω να θεωρείτε ότι τηρήσαμε αυτή τη δέσμευσή μας και χαίρομαι για το έξοχο έργο που πετεθεί. Η μόνιμη ομάδα του ΑΕΦΡΕΣ είπε την προεδρία του Τίοντορ Στολογιάν. Ε, καταρχάς θα αναφερθώ σε τρία βασικά θέματα τι κάνει το ΕΦΡΑΚ τώρα, τα βασικά θέματα, το FRS 17 και θα μιλήσω επίσης και για το FRS 9, ε, το Equity Instrument, τα μέσα αυτά που εξετάζουμε κατά τίμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να καλύψουμε και τις ε, επιθυμίες του Κοινοβουλίου. Το βασικό θέμα. Το μηχάνημα. Διαφάνεια 4 παρακαλώ. Λοιπόν, το FRAG εξετέλεσε μία αποστολή κοινοφελή να εξυπηρετήσει το δημόσιο συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ενώσεως μέσω της επεξεργασίας και πρόθεσης του ευρωπαϊκού οράματος όσον αφορά τις ε, πληροφορίες που δίδονται στον αυτά τα χρηματοστατικά. Οι δραστηριότητε είναι η επιρροή όσον αφορά την προετοιμασία των προδιαγραφών IFRS, τη γνωμοδότηση που βάλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά την έγκριση και τέλος ε, την ε, επίτευξη έρευνας η έρευνα του ΕΦΡΑΓ συμβάλλει στο να δώσει επιφανή θέση στην Ευρώπη στι διεθνεί συζητήσει για τι πληροφορίε οικονομικού περιεχομένου. Το πρόγραμμα το ερευνητικό, τα πρόγραμματα ερευνητικά τα επεξεργάζονται κατόπιν των προδιαγραφών που τίθεται, αλλά και εν συνεχεία διαβούλευση δημόσια που λαμβάνει η χώρα για τον εντοπισμό των προτεραιοτήτων μα. Το ΕΦΡΑΓ σημείωσε πρόοδο, αλλά πάντα μπορούμε να τελειοποιηθούμε και γι' αυτό το 2017 αναθέσαμε σε εξάρτητο φορέα έναν έλεγχο και τα αποτελέσματα είναι γενικώ θετικά και δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα μας και θα τα λάβουμε υπόψη ε, δεόντως στη διαμόρφωση στρατηγικής μας. Εξάλλου το ΕΦΡΑΓ ε, τους επόμενους μήνες θα παίξει το ρόλο του στο σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη χρηματοδότηση της βιώσιμης ανάπτυξης και το ΕΒΡΑΚ, είναι σημαντικό αυτό, θα επίσης θα, είναι, θα υποστηριχθεί από το European ε, Reporting Club. Λοιπόν, τώρα, σημείο αναφοράς στο IFRS 17 είναι αποτέλεσμα 20 ετών προσπαθειών. Θα αντικαταστήσει τα πρότυπα FRS 4 που θεσπίστηκαν το 2004 και επιβαλόταν η μετροποποίησή τους. Το FRS 4 συνελήφθη ως μια προσωρινή λύση που θα επέτρεπε μεγάλη ποικιλομορφία των λογιστικών πρακτικών και αυτό είχε σαν πρόβλημα να δυσχεραίνει τη συγκρισιμότητα των αριθμητικών στοιχείων. Θέλαμε λοιπόν να καλύψουμε τις επιθυμίες των επενδυτών για καλύτερη συγκρισιμότητα χάρη σε μια βελτίωση των λογιστικών πρακτικών που θα ακολουθούνται. Αντίκτυπος της εφαρμογής των νέων προδιαγραφών θα είναι ποικιλόμορφος ανάλογα με τις επιχειρήσεις συναρτήσει των σημαντικών διαφορών που υπάρχουν όσον αφορά τις παρούσες λογιστικές πρακτικές που εμπνέονται από τις εθνικές προδιαγραφές ε, κυρίως στα διάφορα κράτη-μέλη. Πολλές επιχειρήσεις ασφαλιστικές θα επηρεαστούν από τις νέες ε, προδιαγραφές. Το IFRS 17 ε, θα αποτελέσει θα, σημαντική αλλαγή για τον ασφαλιστικό τομέα και εφαρμογή αυτών των διαγραφών συνεπάγεται σημαντικές επενδύσεις ε, σε χρήμα και σε ε, χρόνο. Βλέπετε στην οθόνη το χρονοδιάγραμμα των εργασιών που έχει καθοριστεί και στο τέλος ε, το ΕΦΡΑΓ θα έχει γνωμοδοτήσει βασιζόμενο σε πολύ ε, σημαντική ανάλυση αντιχτύπου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας έδωσε περισσότερο χρονικό περιθώριο από ό,τι είχαμε για τα προηγούμενα πρότυπα. Θα έχουμε έτοιμη την γνωμοδότηση για το τέλος του έτους με δημοσίευση ενός σχεδίου γνωμοδοτήσεως το Σεπτέμβριο και έτσι θα επιτραπεί μια δημόσια διαβούλευση και θα λάβουν χώρα οι εργασίες αυτές και κατά τη διάρκεια της θερινής περίοδου. Ε, ποια εγχειρήματα ακολουθούνται ε, στα πλαίσια του προβληματισμού για τι περιγραφε IFRS 17 το Διοικητικό Συμβούλιο μέσω διαφόρων φορέων, ασφαλιστών, επενδυτών και άλλων συμμετεχόντων ε, άκουσε τις ανησυχίες όλων αυτών των εκπροσώπων ε, που, που προωθήθηκαν. Μελέτη αντιχτύπου ε, μέσω δειγματολογίου ασφαλιστών είναι κάτι που πραγματοποιήθηκε, ξεκίνησε μάλλον, έχει δρομολογηθεί και συνεχίζεται και είτε θα είναι πλήρης ε, η μελέτη δικτύπου είτε θα απλουστευμένη μορφή διοργανώνουμε και προγράμματα διαθρωμένων συνεντεύξεων με τους χρήστες ε, των ε, διαφόρων φορέων στις διάφορες χώρες. Λοιπόν, λοιπόν, καθορίζουμε μαζί με τη Συμβολή Πανεπιστημιακών τα διάφορα θέματα που εξετάζονται και έτσι θα έχουμε μια οικονομική ανεξάρτητη μελέτη που θα εξετάζει τις συνέπειες για τον τομέα, τον ασφαλιστικό στην Ευρώπη, ε, είναι κάτι που έχουμε παραγγείλει, έγινε αυτή η μελέτη, έχουμε αναθέσει. Τώρα, στον προβληματισμό στα πλαίσια του ΕΦΡΑΚ, μετά την έκθεση Μάιστατ, το σημαντικό ήταν να γίνει μια εκτίμηση του ε, European Public Good. Ε, προβληματισμός λαμβάνει υπόψη μελέτη αντιχτύπου που θα εξετάσει τον κίνδυνο για ανεπιθύμητες συνέπειες όσον αφορά τα χρηματοστικά. Ε, πολιτική των επενδύσεων των ασφαλιστών λαμβάνεται υπόψη, οι μακροπρόθεσμες επενδύσεις, η πολιτική των προϊόντων και η τιμολόγηση, η δεσμολόγηση αυτών, η χρηματοστατική σταθερότητα και η ανταγωνιστικότητα του τομέα αυτού του ασφαλιστικού στην Ευρώπη. Έχουμε πλήρη επίγνωση της σημασίας που έχει ο τομέας ο ασφαλιστικός σαν επενδυτή στην ευρωπαϊκή οικονομία, ασφαλιστικό τομέα και σαν πάροχο προστασία για του πολίτε και για τον επιχειρηματικό κόσμο. Και γι' αυτό η εκτίμηση συγκρισιμότητα στα FRS 17 με το European Public Good είναι στο επίκεντρο των εργασιών των προσπαθειών. Και στο τέλος της αναλύσεως θα πρέπει να δούμε κατά πόσο τα φέλη που απορρέουν από την εφαρμογή του FRS 17 είναι ή όχι ανώτερα από το κόστος που θα επιφέρει η εφαρμογή του συστήματος και όσον αφορά τα ποσοτικά στοιχεία και όσον αφορά τα ποιοτικά στοιχεία. Πέρα λοιπόν από αυτή την αξιολόγηση του European Public Good προβαίνουμε και σε αξιολόγηση τεχνικής φύσεως. Οι τεχνικές ε, πτυχές ε, λαμβάνονται υπόψη. Ποιες είναι αυτές. Είναι το επίπεδο λεπτομέρειας, συσχετισμός με το, το επιχειρηματικό μοντέλο του ασφαλιστού, η αναγνώριση του κέρδους, οι μεταβατικές επιλογές και ε, λογιστικό έλεγχο τη αντασφάλιση και των συμβάσεων ειδικών. Ε, εξακριβώνουμε κατά πόσο ε, αντιστοιχούν στα κριτήρια προδιαγραφέ που έχουν εγκριθεί και να δούμε αν οι πληροφορίε που παράγονται είναι ειλικρινεί και αξιόπιστε και ακολουθούν συνετή προσέγγιση. Διάφοροι θεωρούν ότι το FRS 17 οδηγεί σημαντική πρόοδο όσον αφορά τι οικονομικέ πληροφορίε και παραμένουν διάφορα θέματα που χρειάζονται περαιτέρω και ενδελεχέστερη ανάλυση. Ινδού λοιπόν τα βασικά στοιχεία που ήθελα να αναφέρω για τα FRS 17. Προφανώς η συζήτηση θα μας επιτρέψει να προβούμε σε λεπτομερέστερη εξέταση και να δώσουμε απαντήσεις σε ερωτήσεις σας με την αποτελεσματική συνεργασία που θα έχουμε όσον αφορά τα τεχνικά ζητήματα, όταν είναι πολυτεχνικής φύσεως να σας πω κάποια πράγματα για τον προβληματισμό των παρόντων για το FRS 9 ε, και το Liquidity Instruments. Λοιπόν, στον προβληματισμό για το FRS 9 τον Οκτώβριο του 2016 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι το FRS 9 θα ήταν θετικό όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Στατηγική των Μακροπρόθεσμων Επενδύσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από το ΕΦΡΑΚ να γνωμοδοτήσει επ' αυτού. Η πρώτη φάση ήταν σχετικά δύσκολη αφορούσε τη συλλογή ε, πληροφοριών και επιπλέον είχαμε άλλη μια δυσκολία να διατυπώσουμε ορισμούς των μακροπρόθεσμων αυτών επενδύσεων. Τι αποτελεί μακροπρόθεσμη επένδυση. δεύτερη φάση, να προσπαθήσουμε να βρούμε ενδεχόμενες λύσεις επικεντρωνόμενοι επί των δυνατοτήτων να επιτρέψουμε μια ανακύκλωση αν αυτή είναι πλαισιωμένη. Ε, έχει δρομολογηθεί μέχρι τέλος ε, μήνα Μαΐου ο προβληματισμός και οι συζητήσεις για να ακούσουμε τις απόψεις των εμπλεκομένων μερών. Ελπίζει η ΕΦΡΑΚ να προβεί σε συστάσεις ε, το τρίτο τρίμηνο ενεστώτος έτους. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Είμαστε στη διάθεσή σας για να δώσουμε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας. Thank Σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν πάρα πολύ σφαιρική και πλήρης η παρουσίαση. Ο κύριος Στόμιγιαν έχει ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς ορίσατε κύριε Γκοζέ. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας βλέπουμε στη συνάντηση της ΕΚΟΝ. Θα ήθελα να υπενθυμίσω στους συναδέλφους πως τα τελευταία πιο πρόσφατα χρόνια είχαμε τρία πρότυπα τα οποία με το δικό τους τρόπο θα αλλάξουν το επιχειρηματικό μοντέλο στο χρηματοδοτικό κλάδο. Μιλάμε για το IFRS 16 που είναι το leasing, το 9 που είναι τα χρηματοπιστωτικά εργαλεία και τώρα αντιμετωπίζουμε και το IFRS 17 που έχει να κάνει με τα ασφαλιστήρια. Διαβάσαμε ε, τα έγγραφα τα οποία μας στείλατε εσείς και πρέπει να πω πως για τις ασφαλιστικές εταιρείες το 17 είναι πολύ πιο περίπλοκο από το IFRS 9 που καλύπτει τον τραπεζικό κλάδο και τις επιχειρήσεις εκεί. Γιατί? Γιατί μια ασφαλιστική εταιρεία θα πρέπει να ε, εφαρμόσει το 9 για το κομμάτι των στοιχείων ενεργητικού και για τις επενδύσεις που κάνουν και το 17 ε, για τις ε, ευθύνες. Το οποίο σημαίνει ότι είναι εξαιρετικά περίπλοκο να ανταποκριθούν στις απαιτήσει όλων αυτών των νέων προτύπων και κανόνων. Ρωτώ λοιπόν τα εξής. Και η πρώτη μου ερώτηση είναι έχουμε κάποια ενημέρωση για το τι συνέβη σε επίπεδο ασφαλιστικών εταιριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί οι ασφαλιστικές εταιρείες είχαν την δυνατότητα να καθυστερήσουν την εφαρμογή του 9 μέχρι την 1η Ιανουαρίου του 2021, όπου ε, υποτίθεται πως θα εφαρμοστεί και το 17. Δεύτερον, Σύμφωνα με τα στοιχεία που μας ε, έστειλε η ICB, το IFRS 17 δεν θα έχει επιπτώσεις στην ασφαλιστική αγορά, τουλάχιστον σε επίπεδο διαφοροποίησης ασφαλιστικών προϊόντων ή ε, στις ε, τιμές των προϊόντων αυτών. Εσείς τι νομίζετε σε αυτή τη φάση που βρίσκεται. Τρίτον, για το πόσο περίπλοκη θα είναι η εφαρμογή του IFRS 17 και το πώς θα το κάνουν αυτό οι ασφαλιστικές εταιρείες. Τα μηνύματα που λάβαμε ήταν πως είναι θέμα χρόνου. Είναι θέμα κόστους και είναι και θέμα επανεκπαίδευσης για πολλούς από τους εμπειρογνώμονες που εργάζονται στον κλάδο αυτό. Ποιος θα τα κάνει όλα αυτά. Σαφέστατα η πρώτη ευθύνη βαρύνει τις ασφαλιστικές εταιρείες. Αλλά η ΕΦΡΑΚ και η ICB τι μπορούν να κάνουν για να βοηθήσουν τις εταιρείες αυτές και ποιος θα παρακολουθεί το τι γίνεται και το κατά πόσο αυτές οι ασφαλιστικές εταιρείε θα εφαρμόσουν κατάλληλα και στον, χρόνο που χρειάζεται αυτά τα νέα πρότυπα και κυρίως το 17. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητέ φίλε, Τεοντόρ. Πολύ καλές ερωτήσεις και επειδή είμαι πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ε, του οργάνου αυτού, φροντίζω να έχουμε στενές σχέσεις με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και να ακούμε όλες τις απόψεις. Για το τεχνικό σκέλος ακόμα κάποια στοιχεία πρέπει να συμπληρώσουμε. Αλλά θέλω να δώσω μία απάντηση σε όλα από τα θέματα τα οποία έθεσες για την ε, εμπειρία που είχαμε από τις επαφές μας με ασφαλιστές ή επενδυτές. για τη διαφορά μεταξύ του προτύπου 9 και την εφαρμογή αυτού και την τροπολογία ε, που εγκρίθηκε σε αυτά και τα οποία ε, ε, επεκτάθηκαν και στις ασφαλιστικές τράπεζες, να σας πω πως είμαστε σε επαφή με μια σημαντική εταιρεία η οποία υπολόγισε το εξής, ότι με το πρότυπο 9 αν είχε εφαρμοστεί συνέχεια και με την εφαρμογή του διαφοροποιημένου ουσιαστικά καταλήγουμε σε διαφορετικά αποτελέσματα, σε διαφορετικά επίπεδα επιπτώσεων, αλλά δεν έχω τα αριθμητικά στοιχεία για τα δύο σενάρια που περιμένω τις επόμενες εβδομάδες. Τώρα, πώς θα επηρεαστεί η αγορά. Αυτή τη στιγμή οι ασφαλιστές δεν επιμένουν στο σημείο αυτό. Η επιπτωσιολογική μελέτη θα γίνει και όταν γίνει ίσως θα έχουμε την απάντηση. Αντίθετα, απαιτούν να λάβουμε υπόψη το πόσο περίπλοκος είναι ο μηχανισμός και πως το ότι χρειάζονται ε, επαρκή μέσα και πόροι για να εφαρμοστεί το πρότυπο 17 για το οποίο δεν έχουν ουσιαστικές αντιρρήσεις. Δεν έχουμε δηλαδή επικρίσεις για το ίδιο το πρότυπο, αλλά οι ανησυχίες τους έχουν να κάνουν με τις συνθήκες εφαρμογής αυτού του προτύπου, το κόστος της εφαρμογής, όπως επίσης και την ύπαρξη ανθρώπινων πόρων που θα επιτρέψουν να κάνουμε τη σημαντική αυτή προσπάθεια που γίνεται για να εφαρμοστεί. Αυτά είναι λοιπόν τα στοιχεία στα οποία θα πρέπει να σκεφτούμε ε, σε σχέση με τις παρατηρήσεις που έχουν γίνει και τα όσα θα μας πούνε και να σας πω πως γύρω στις, νομίζω στις 3 Ιουλίου θα συναντηθούμε με ασφαλιστές και αντασφαλιστές, οι οποίοι σίγουρα θα συμπληρώσουν και θα διευκρινίσουν αυτή την επιστολή την οποία λάβατε και εσείς και εμείς από, την, από το φόρουμ, που περιγράφει τις ανησυχίες, δεν θα έλεγα τις αντιρρήσεις, τις ανησυχίες για το χρόνο εφαρμογής και για το χρόνο που είναι απαραίτητος για την εκπαίδευση του αρμοδίου προσωπικού. Δεν ξέρω αν ο συνάδελφος θέλει να συμπληρώσει κάτι. Ελπίζω να έχω απαντήσει σε αυτά που ρώτησες. Ευχαριστώ. Θέλετε να συμπληρώσετε κάτι. Όχι, όχι. Νομίζω ότι ο Ζαν Πολ τα κάλυψε όλα. Η κυρία Μπερέζα. Ευχαριστώ αγαπητέ Πρόεδρε. Αγαπητέ συνάδελφοι και φίλοι, αγαπητέ Ζων Πολ. Κάτι που δεν αναφέρθηκε ακόμη σε αυτή τη συζήτηση είναι η σημασία που ελπίζω να αποδώσετε στο ψήφισμα που εκπονεί τώρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και που θα εγκριθεί κατά την Ολομέλεια του Ιουλίου. Έχουμε προσαρμόσει το χρονοδιάγραμμά μας ε, με βάση τις πληροφορίες που μας δίνουν τώρα οι ασφαλιστές για να δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτή η προδιαγραφή. Όλοι θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξει, αλλά τώρα πρέπει να δούμε και τις λεπτομέρειες. Οπότε, πρώτα απ' όλα, σε τι επίπεδο θα αθρίζονται οι κίνδυνοι με βάση αυτή τη νέα νόρμα μήπως ε, θα μειωθούν οι πληροφορίες που θα είναι διαθέσιμες και ανταποκρίνεται στα χαρακτηριστικά των συμβολέων που μας δίδουν οι ίδιοι ασφαλιστές. Δεύτερη ερώτηση, την αναφέρατε κάπως όταν συζητήσαμε το IFRS 9. Τις τράπεζες που επίσης έχουν ε, και ασφαλιστικές λειτουργίες ποια θα είναι η συμβατότητα μεταξύ των IFRS 9 και 17. Επίσης, πολλοί ενδιαφερόμενοι ανησυχούν, αν και άλλοι όχι, για το κόστος ε, της εφαρμογής αυτής της νέας νόρμας σε σχέση με το όφελος που θα αποκομίσουν. Πώς θα αντιμετωπίσετε τα επιχειρήματα αυτά, γιατί κάποιοι θα τα θέσουν. Ως πρόεδρος του ΕΦΡΑΓ να σας θέσω άλλη μία ερώτηση, πιο γενική. Πώς αξιολογείτε το ρόλο που παίζουν αυτές οι νόρμες, οι λογιστικές νόρμες. Για να αξιολογηθεί λοιπόν σωστά η υγεία των επιχειρήσεων, γιατί η ψηφιοποίηση ε, δημιουργεί νέες καταστάσεις που δεν λαμβάνουν την υπόψη από, αυτές τις, ε, από αυτά τα λογιστικά πρότυπα. Υπάρχουν λοιπόν πολλά δεδομένα που δεν τα λαμβάνουν υπόψη τα λογιστικά πρότυπα, τα οποία υποτίθεται ότι πρέπει να περιγράφουν σωστά και να μας παρουσιάζουν σωστά την κατάσταση των επιχειρήσεων. Πώς λοιπόν θα λάβετε υπόψη αυτά τα νέα στοιχεία που παίζουν ρόλο τελικά στην κατάσταση και την υγεία των επιχειρήσεων. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε για αυτές ε, τις ερωτήσεις. Δεν θα απαντήσω στα τεχνικά θέματα. Για το επίπεδο άθρησης ε, των στοιχείων. Από ό,τι καταλαβαίνω η κύρια ανησυχία των ασφαλιστών, των ασφαλιστικών εταιριών είναι ότι ο κίνδυνος δεν είναι ε, ότι δεν θα καταλαβαίνουμε πώς λειτουργούν οι επιχειρήσεις, αλλά ότι δεν θα επιτρέπεται η αμοιβεοποίηση. Η Άξα το τόνισε αυτό. Για τις τράπεζες που λειτουργούν και ως ασφαλιστικές, σήμερα είναι ικανοποιημένε που έχουν δυνατότητα να εξαιρεθούν από την προδιαγραφή και το ΕΦΡΑΚ έπαιξε πραγματικό ρόλο σε αυτό γιατί με βάση την παρατήρηση που περιεχόταν στην νομοδότησή μας για το ενδεχόμενο του ανταγωνισμού με βάση αυτό η Επιτροπή και τα κράτη-μέλη διεύρυναν ε, την ε, τροπολογία για το IFRS 4 Τώρα για το κόστος σε σχέση με το όφελος. Καταλαβαίνω την ανησυχία σας γιατί τη συμμερίζομαι. Να μιλήσω τώρα προσωπικά. Αν εξετάσουμε, έχουμε την εντύπωση ότι άλλοι θα φέρουν το κόστος και άλλοι θα δρέψουν το ωφέλη. Γιατί το κόστος θα είναι των ασφαλιστών που θα πρέπει να συμμορφωθούν και το όφελος, το κέρδος θα το πάρουν οι επενδυτές γιατί θα γνωρίζουν την κατάσταση των επιχειρήσεων και άρα θα επενδύσουν σωστά. Αυτή είναι μια πλευρά που θα πρέπει να μελετήσει η μελέτη αντικτύπου για να καθορίσουμε πολύ σωστά την κατάσταση. Για παράδειγμα, μια μεγάλη βρετανική εταιρεία, οι βρετανικές εταιρείες γενικά είναι ευνοϊκές προς, το προς τα IFRS, μια βρετανική εταιρεία τονίζει ότι θα είναι τεράστιο το κόστος της εφαρμογής αυτής, ε, αυτού του νέου προτύπου για το τελευταίο που είπατε ότι πρέπει να έχουμε και περαιτέρω στοιχεία σε αυτά μας τα πρότυπα. Ναι, το καταλαβαίνουμε. Και αυτός ο έλεγχος που ανέφερα προηγουμένως το λέει και αυτό, ότι πρέπει να διευρύνουμε δηλαδή τα δεδομένα που λαμβάνουμε υπόψη και τα κριτήρια. Αλλά εμείς ως Εφράγκα είμαστε απλώς η βάση επί του οποίου βασίζεται το ΛΑΜΠ για να συλλέξει στοιχεία για τις επιχειρήσεις. Αυτό θα επιτρέψει να διευρύνουμε τα στοιχεία και τα κριτήρια χωρίς να έχουμε περιορισμούς. Γιατί πρώτα θα σκεφτούμε. Θα υπάρχουν κάποιες ομάδες εργασίας. Αλλά δεν μπορώ να σας πω κάτι πιο συγκεκριμένο. Η Κομισιόν θα μας υποβάλει ένα οδικό χάρτη για να διευρύνουμε την συζήτηση. Και τώρα ο Άντζο. Ευχαριστώ. Το επίπεδο εφαρμογής είναι από τα βασικά θέματα που εξετάζει η ΕΦΡΑΚ. Όπως σε πολλούς τομείς υποβολής στοιχείων οικονομικών υπάρχει και ένα αντάλλαγμα πολύ ψηλό επίπεδο ομαδοποίησης ίσως να ταιριάζει περισσότερο με κάποιες αξιολογήσεις κινδύνου και κάποιες τιμολογήσει και τι σχετικέ αποφάσεις στον τομέα, αλλά αυτό το πολύ ψηλό επίπεδο ομαδοποίηση μπορεί να καλύπτει και διάφορες τάσει στην κερδοφορία προϊόντων που κάποιοι επενδυτέ θεωρούν ότι είναι χρήσιμο, οπότε αυτό είναι ένα κομμάτι τη αξιολογήσεω. Βασικό στοιχείο ε, ε, λοιπόν, και έχει χρειάζεται ένα συγκεκριμένο έγγραφο για να ευαισθητοποιηθούν οι εμπλεκόμενοι φορεί. Όσον αφορά την κατά περίπτωση εφαρμογή, ε, εγώ το προβλέπω ότι η ΕΦΡΑΚ θα μπορέσει να, υπό κάποιου συγκεκριμένου όρου να μπορέσει να εκτιμήσει το κόστος εφαρμογής αλλά ε, περισσότερο ποιοτική φύση θα έχει αξιολόγηση του όφελους, το φέλους. Αυτό είναι γνωστό στι αξιολογήσει συνεπειών. Οπότε το πρόβλημα για του ευρωπαϊκού θεσμού και για την ΕΦΡΑΚ θα είναι η εξισορρόπηση μεταξύ ποσοτικοποιημένων στοιχείων και ποιοτικών στοιχείων. Τέλος, όσον αφορά την ψηφιακή οικονομία, ε, μία από τις μελλοντικέ έρευνες που θα κάνει η ΕΦΡΑΚ θα είναι για τα κρυπτο στοιχεία ενεργητικού, ας τα αποκαλέσω έτσι, θα δούμε κατά πόσο οι εμπλεκόμενοι φορείς θα στηρίξουν ένα τέτοιο εγχείρημα στα πλαίσια το, της αναφοράς στοιχείων για τα οικονομικά. Με έτσι, έτσι που εξελίσσονται οι οικονομίες μας και έχουν περισσότερο εξάρτηση σε άειλα προϊόντα, οι περισσότερες προσπάθειες θα γίνουν για ενημέρωση θα, είναι, ε, θα διαφοροποιηθεί. θα βασιστούμε και στο εργαστήριο που ανέφερε ο Ζαν Πολ. Είναι κρισίμου σημασία η συνδρομή του όσον αφορά την προσέγγιση μα ε, για, αυτά τα, για την ενημέρωση αυτά τα καινούργια στοιχεία. Ευχαριστώ, κύριο Καμάλ. Ευχαριστώ, χαίρομαι που σε βλέπω, Ζαν Πολ. Απόλαυσα πρώτερε σύντομε κουβέντε που είχαμε στα αγγλικά. Λοιπόν, Μία-δύο ερωτήσει έχω. Που απορρέουν από αυτά που ηθήκησαν προ... προηγουμένω. Θα θυμόσαστε ότι δημιουργήσαμε την ομάδα εργασία στο ΕΦΑΡ στο Κοινοβούλιο, διότι υπήρχαν ανησυχίε για τα αποτελέσματα τη οικονομική κρίση. Εγώ πάντα είχα τρία προβλήματα. Τον ήταν τράπεζε μου έλεγαν ότι είναι τράπεζε πολύ μεγάλε για να χρεοκοπήσουν και περιμέναμε να στηριχθούν από του φορολογούμενου. Δεν έχει λυθεί το πρόβλημα, θα το συζητήσουμε. Το δεύτερο, ε, οι διευθυντές, οι ευθύνες των ε, διευθυνών των ε, ε, στελεχών. Ίσως έχουμε προβλήματα τα CDR και CDS. Υπάρχουν κάποιοι διευθυντές τραπεζών που είναι υπερφύαλοι στην προσέγγιση τους γι' αυτό. Ήμουν σε μια εκδήλωση της προάλλας και ένας διευθυντής τράπεζας μου είπε ότι είναι διευθυντής. Και ήταν πολύ αλαζονικός στη συμπεριφορά του. Μετά από την κρίση έρχεται ένας τύπος λοιπόν από την HSBC και έλεγε ότι είναι διευθυντή και ήταν φοβερά λαζονικό. και έπρεπε να είναι πιο ταπεινόφρον. Αυτό θεωρώ. Τρίτον, είναι τα λογιστικά πρότυπα. Η συζήτηση τότε αφορούσε προβλέψεις για δάνεια με διαβίου διάρκεια, αναμενόμενες και απροσδόκητες απώλειες, οι απροσδόκητες πώς καλύπτονται, πώς εξασφαλίζονται οι τράπεζες ότι ε, χρησιμοποιούν, εκδίδουν χρηματοστατικά ε, χρηματοδοτικούς τίτλους χωρίς να καλύπτουν ενδεχόμενες ε, απώλειες. Τι γίνεται με τις απροσδόκητες απώλειες, πώς τις καλύπτεται. Έχω μια-δύο ερωτήσεις. Η πρώτη. Τότε επικρίναμε την ΕΦΡΑΓ και θα ήθελα να ξέρω πώς βλέπετε εσείς τον έλεγχο Πού, πάει καλά η ΕΦΡΑΓ, αλλά πού πρέπει να βελτιωθεί η ΕΦΡΑΓ για να έχουμε εμεί μεγαλύτερη εμπιστοσύνη απέναντί σα. Συλλογικά συμφωνούμε ότι η ΕΦΡΑΚ έχει βελτιωθεί και χάρη στην ε, ηγεσία σας. Τι, πού μπορεί να βελτιωθεί όμως περισσότερο. Δεύτερον, IFRS 17. Κάποιες ε, χώρες, κάποιες εταιρείες διαμαρτύρονται γι' αυτό. Μας δίνετε κάποια γεύση. Περί τίνος πρόκειται λόγω επιχειρηματικών μοντέλων σε κάποιες χώρες. Ποιες χώρες είναι αυτές που διαμαρτύρονται. Ποιες είναι αυτές που είναι ικανοποιημένες διότι δεν επηρεάζεται πολύ το επιχειρηματικό τους μοντέλο. Δεν θέλω να δώσω πολιτική απόψη αυτά που λέω. Ποιες χώρες είναι ικανοποιημένε με τα FRS 17 και ποιες ανησυχούν οι ασφαλιστές τους. Γιατί αναφερθήκατε, είπατε ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα όσον αφορά ασφαλιστέ από κάποιε χώρε. Αυτό θα ήθελα κάποια διευκρίνηση. Ευχαριστώ. Είναι η απάντηση. Ξεκινάει η απάντηση μάλλον. Θα απαντήσω γαλλιστή. Τώρα όσον αφορά το σχόλιο σας για τον έλεγχο ε, αντίληψη, σύλληψη αν θέλετε να πω ότι τα αποτελέσματα ήταν θετικά όσον αφορά το επίπεδο ικανοποίησης. Επί ευκαιρία του ελέγχου αυτού διαπιστώσαμε ότι υπήρχαν συμπληρωματικές απαιτήσεις και πληροφορίες. Και ο ρόλος που παίζει το ΕΦΡΑΓ όσον αφορά το πώς επηρεάζει τις προδιαγραφές IFRS πριν ολοκληρωθούν, αυτό δεν γίνεται απόλυτα αντιληπτό τι ρόλο παίζουμε. Ε, με τρόπο πολύ διακριτικό εργαζόμεθα. Και έτσι το ουσιαστικό έργο που γίνεται τις ομάδες και από την ομάδα τεχνικών εμπειρογνωμόνων ή από τις ομάδες εργασίες, οι εργασίες αυτές δεν γίνονται επαρκώς αντιληπτές παρόλο που προβάλλονται στην ιστοσελίδα μας και όλες οι εργασίες της έφραγκ είναι απόλυτα διαφανείς, διότι όλα τα κείμενα δημοσιεύονται, τα σχόλια, οι επιστολές εμφανίζονται στην ιστοσελίδα μας στο διαδίκτυο που είναι προσβάσιμη σε όλους. Είναι μια προσπάθεια πράγματι που πρέπει να γίνει από την πλευρά μου από όταν είμαι πρόεδρος προσπαθώ να ισχύσω τη σχέση με το Κοινοβούλιο. Απόδειξη αυτού σήμερα. Ποτέ πριν δεν υπήρξε άμεση επαφή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ακόμα και αν υπήρχαν καρποφόρες επαφής με το FRS Team. Βασιζόμαστε σε ενίσχυση των εργασιών και να γίνουν όλα πιο ορατά. Να ακουγόμαστε περισσότερο. Πιστεύω ότι σύντομα, στο εγγύς μέλλον, ο ρόλος των βουλευτών θα μας τροφοδοτήσει τον προβληματισμό μας. Από αυτή την πλευρά σας διαβεβαιώνω, κυρία Πρόεδρε, κυρία Μπερές, θα διαβάσουμε με τα προσοχής και όχι μόνο με τα προσοχής διαβάσουμε, θα λάβουμε υπόψη μας όλο όσον αφορά που θα ήθελε να εκφράσει στο ψήφισμά του το Κοινοβούλιο. Όσον αφορά τους ικανοποιημένους και μη ικανοποιημένους, τις χώρες που είναι ικανοποιημένες και αυτές που δεν είναι. Είναι περισσότερες οι αποχρώσεις. Εν γέννη υπάρχει μια πλειοψηφία ε, φορέων που λέει ότι οι προδιαγραφές είναι χρήσιμες και σκόπιμες. Εγώ θα έλεγα αυτό που ανησυχεί είναι ο περίπλοκος χαρακτήρας εφαρμογής των προδιαγραφών και ενδεχόμενο το κόστος και ανάγκη ανθρωπίνων πόρων που απαιτούνται για την εφαρμογή των προδιαγραφών. Τώρα ε, ζητήσετε χαρτογράφηση των χωρών που είναι υπέρ και ποιε είναι κατά. Δύσκολο να γίνει αυτό. Σύμφωνα με παλιά θεωρία που διαμόρφωσα στο Κοινοβούλιο παλιά, αφορά και τον τρόπο με τον οποίο οι διάφοροι αντιλαμβάνονται το, την εφαρμογή του δικαίου. Όταν είμαστε σε χώρες που έχουν αγγλοσαξονική ε, προσέγγιση στον αφορά το δίκαιο, ε, υπάρχει γενικά ο νόμος και μετά ε, στην εφαρμογή του νόμου γίνεται κατάλληλη εκτίμωση. Στο, στο ρωμαϊκό δίκαιο, στις χώρες που εφαρμόσει το ρωμαϊκό δίκαιο, Χρειάζεται μεγαλύτερη δυνατή νομική ασφάλεια και οι λεπτομέρειες να καθορίζονται. Μπορώ, θα μπορούσα ίσως να πω ένα μικρό λόγο που δύσκολα μεταφραστεί. Έχουν μανία με το κείμενο οι Γάλλοι νομικοί. Θέλουν πάντα περισσότερε διευκρινήσει. Κολλάνε στι λέξει. Και όταν παίρνουν τι ε, βλέπουν του ενοχλούν, ενοχλούν οι διευκρινήσει. Και μετά έχετε άλλο είδο χωρών, όπω είναι οι φίλοι μα οι Γερμανοί. εκεί δεν ικανοποιημένοι με τους κανόνες που υιοθετούνται, αλλά από τη στιγμή που υιοθετούνται οι κανόνες εφαρμόζουν τους κανόνες. Υπάρχει ένα φάσμα λοιπόν συμπεριφορών όσον αφορά την αποδοχή του IFRS 17. Αλλά επιμένω ότι κανείς δεν απορρίπτει αυτές τις προδιαγραφές και γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να βρούμε λύσεις που θα επιτρέψουν χάρη στο έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των διαφόρων ομάδων και επιτροπών ε, να βρούμε λύσεις στα διάφορα κρίσιμα ζητήματα που θα είναι αποδεκτές και δεν θα επηρεάσουν την εφαρμογή των ε, προδιαγραφών. Αυτά και ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ και εσάς για μια πολύ ενδιαφέρουσα αξιολόγηση των νομικών παραδόσεων ε, που έχουμε. Η κυρία Νακτγκάλ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε κοντά μας σήμερα και ήθελα να σας πω πως εκτιμάμε ιδιαίτερα τη δουλειά που κάνετε εσείς και το προσωπικό σας για να αναλύσετε το πώς αυτά τα πρότυπα θα έρθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχω κάποιες ερωτήσεις σχετικά με τις ε, προσθήκες στα ασφαλιστήρια και το πώς αυτό θα συνδυαστεί με τα όσα έχετε στο πρότυπο 17. Καταρχήν, η ημερομηνία εφαρμογής 1η Ιανουαρίου του 2021 πώς σας βρίσκει και επίση η μετάβαση από το παλιό πρότυπο προς το καινούριο πώς θα εξασφαλιστεί πώς θα είναι ομαλή, γιατί δεν είναι εύκολο. Και τι θα γίνει με τον κλάδο των ασφαλιών. Θα μπορέσουν να σεβαστούν και να συμμορφωθούν με τις διατάξεις περί υποβολής αναφορών που έχετε στο πρότυπο και εν ώψη της ημερομηνία εφαρμογή της 1ης Ιανουαρίου του 2021. Επίσης, οι ΙΠΑ δεν συμμετέχουν στο πλαίσιο αυτού του πρότυπου, δυστυχώ κατά τη γνώμη μου, οπότε θα έχουμε αρκετές διαφορές μεταξύ των Αμερικανικών και των Ευρωπαϊκών προτύπων. Οπότε, με ποιο τρόπο έχετε σκοπό εσείς να αντιμετωπίσετε αυτό ε, στην ε, περίπτωση, στο στατικές που μελετάτε εσείς. Χτες η Επιτροπή μας συζήτησε την αναθεώρηση του επίπεδου 2 της Φερεγγιώτας 2. Και την επόμενη εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κάνει και μια γενικότερη αξιολόγηση των κεφαλικών απαιτήσεων για τον κλάδο των ασφαλιών. Έχετε να μας πείτε τι θα γίνει και με τη Φερεγγιότητα 2 και πώς το πρότυπο 17 θα την επηρεάσει και αντίστροφα. Και επίσης, επαναλαμβάνω, μπορείτε να μας ε, αναφέρετε δύο λόγια για την περίπτωση που μελετάτε ως study case. Ευχαριστώ πολύ. Οι ομερμηνίες εφαρμογής που είναι η 1η Ιανουαρίου 2021 είναι ένα θέμα το οποίο προκαλεί όλο και περισσότερες συζητήσεις. Έχουμε 3,5 χρόνια ακόμα μπροστά μας από τη στιγμή της δημοσίευσης του προτύπου και σε σχέση με άλλα μεγάλα πρότυπα νομίζω είναι μια μάλλον γενναιόδορη περίοδος μέχρι την εφαρμογή. Παρ' όλα αυτά προφανώς είναι περίπλοκο, είναι δύσκολο, οπότε όταν κλείσουν οι διάφορες μελέτες περιπτώσεων, ε, οι case studies, θα έχω πιο πολλά να σας πω χτες, Κοίταξα μία έρευνα που έκανε μία ανεξάρτητη, ένας ανεξάρτητος φορέας ιδιωτικού κλάδου και είπε πως 100 μάνετζερ στον, ε, σε, ένα κράτος μέλος και 90 σε ένα άλλο κράτος μέλος από τον τομέα των ασφαλείων είπαν πως θα είναι έτοιμοι. Αλλά εντάξει, αυτό δεν σημαίνει κάτι για μας. Γιατί είπα, όπως είπατε κι εσείς, αποφάσισαν να μην εφαρμόσουν για εγχώρια ε, καταχώρηση το δικό μας πρότυπο. Έχουν το δικό τους σχέδιο που δεν αποτελεί κοινό σχέδιο με τα διεθνή ε, λογιστικά πρότυπα και το σχετικό συμβούλιο, αλλά θα δούμε τι θα γίνει. Νομίζω ότι θα εξελιχθούν προς την ίδια κατεύθυνση με το δικό μας πρότυπο και αυτό που κάνει η ΕΦΡΑΚ αυτή τη στιγμή είναι μια λεπτομερή συγκριτική μελέτη μεταξύ των δικών μας απαιτήσεων και τα βασικά ανταγωνιστικά πλαίσια που είναι αυτά που ισχύουν στη ΣΥΠΑ και στην Ιαπωνία. Είναι μια τεχνική μελέτη αλλά στα πλαίσια της διαβούλευσης που κάνουμε ζητάμε να μας πούν αν υπάρχουν στοιχεία που να οδηγούν ε, σε προβλήματα ανταγωνισμού, πλεονεκτήματα ή μειονεκτήματα, ακριβώς λόγω των διαφορών που έχουμε ε, σε αυτά τα λογιστικά πρότυπα. Για το φερικαιότητα 2 ένα κομμάτι της προσπάθειάς μας έχει να κάνει με την αξιολόγηση ε, των ομοιοτήτων και των διαφορών μεταξύ Φερεγγιώτας 2 και του προτύπου 17. Δεν νομίζω ότι αυτό θα ελαφρύνει το κόστος εφαρμογής του προτύπου, αλλά δεν έχουμε αυτή τη στιγμή μια ε, μελέτη για να ε, συμπεριληφθούμε και εμείς στην μελέτη του Φερεγγιώτα 2 και νομίζω ότι για το πρότυπο 17 δεν ξέρουμε αν θα έρθουν πιο κοντά ή θα απομακρυνθούν, αλλά νομίζω ότι και αυτό ε, θα φανεί μετά από το τέλος των μελετών που θα γίνουν. Μια διευκρίνηση για την διεθνή και αμερικανική πτυχή. Πρόσφατα ε, συνάντησα την, τον πρόεδρο της Ίγκον, μια ασφαλιστική εταιρεία ε, που έχει έδραση στις κάτω χώρες και έχει μεγάλη διεθνή δράση και συζητήσαμε το θέμα του ανταγωνισμού με τη ΣΥΠΑ και θα κάνουμε και μία τεχνική συνάντηση μαζί του στις 19 ε, Ιουνίου με τον Άντριο στις Βρυξέλλες και με τους τεχνικούς τους διευθυντές για να μας δώσουν ε, στοιχεία για να τα μελετήσουμε. Έτσι ε, εργαζόμαστε. Δεν ε, δεχόμαστε ότι μας λένε τα λόμπια, αλλά τους ακούμε και κάνουμε κάποιες τεχνικές συζητήσεις για να συζητήσουμε θέματα που τους ανησυχούν με τους πραγματογνώμενες που θα μας βοηθήσουν. Η ΆΕΦΡΑΚ δεν είναι ε, νομοθέτης προτύπων. Εμείς είμαστε συμβουλευτικό όργανο για μια σειρά κανόνων που εγκρίνονται έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Ένωση να δουν κατά πόσο χρήζουν εφαρμογής και κατά πόσο είναι ε, συνεκτικοί με τους περιορισμούς που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Ευχαριστώ, ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος, κυρία Ματίας. Ευχαριστώ και καλώς ήρθατε πίσω στο σώμα στο οποίο συμμετείχατε. Δύο πολύ συγκεκριμένες ερωτήσεις για τις πρόσβατες, πρόσφατες δραστηριότητες του ΕΦΡΑΓ. Γιατί πρόσφατα υπήρχε μια συνδιάσκεψη για την σωστή αξία και τέθησαν ε, πολλές ενδιαφέρουσες ερωτήσεις στο πλαίσιο αυτό. Ήθελα να μάθω λοιπόν εάν η ΕΦΡΑΓ θέλει να ασχοληθεί με την προκυκλική φύση της δίκαιης αξίας. Υπάρχει οικονομική ανάκαμψη τώρα, λόγω της νομισματικής πολιτικής. Αλλά, δυστυχώς, και κατά τη γνώμη μου, γιατί δεν είναι σωστό το μείγμα πολιτικών, παρατηρούμε επίσης αυξανόμενες ανησυχίες γιατί σε κάποιους τομείς οικονομικής δραστηριότητας μοιάζει να ξαναξεκινάνε φούσκες. Θέλω να μάθω λοιπόν εάν η ΕΦΡΑΚ θέλει να κάνει μια οικονομική ανάλυση για να συμβάλλει στην αποφυγή αυτών ε, της δημιουργίας ε, τέτοιων φουσκών. Ε, επίσης, για το θέμα της βιώσιμης ανάπτυξης. Ξέρω το θέμα είναι επίμαχο, ότι πολλές συζητήσεις γίνονται, αλλά προκύπτουν ορισμένα θέματα και θα ήθελα να μου πείτε, εάν είναι δυνατόν, να μας πείτε ποια είναι η θέση σας, λαμβάνοντας ε, και να μας πείτε τι συζητήσεις κάνετε για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια και εγώ χαίρομαι που σας ξαναβλέπω. Πολύ τεχνικές ερωτήσεις. Θα απαντήσει ο Άντρου. Είμαστε ομάδα. Ο ένας είναι ο τεχνικός εμπειρογνώμων και εγώ είμαι ο άλλος. Αλλά αναφερθήκατε σε μια συνεδρίαση που έγινε στις 5 Δεκεμβρίου για την fair value, την ε, δίκαιη αξία, όπου νομίζω ότι αναφέρθηκαν πολύ ενδιαφέρουσε ιδέες. Γνωρίζω αυτό το πρόβλημα της προκυκλικότητας γιατί έπαιξε ρόλο στην κρίση. Αλλά για τις λεπτομέρειες να δώσω το λόγο στον Άντζου. Ευχαριστώ. Να απαντήσω όσο μπορώ για τη δίκαιη αξία. Η ΕΦΡΑΓΚ στα πλαίσια του σχεδίου δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την βιώσιμη χρηματοδότηση θέλουμε να δούμε αν υπάρχουν διαφορετικές μέθοδοι μέτρησης των επενδύσεων σε αξιόγραφα πέρα από την δίκαια αξία. Δεν έχουμε ακόμη λάβει επίσημο αίτημα για να κάνουμε κάτι τέτοιο, αλλά όταν υποβληθεί θα το εξετάσουμε. Γενικά. Η διάσκεψή μας ε, στις 5 Δεκεμβρίου κατέληξε σε πορίσματα που είναι δημόσια. Αλλά αυτό που μας λένε και οι πανεπιστημιακοί όλο και πιο συχνά είναι ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία ότι έπαιξε ρόλο ο, στην κρίση η λογιστική αντιμετώπιση ε, που λάμβανε υπόψη την δίκαια αξία. Αλλά μέχρι στιγμής ε, έτσι έχουν τα πράγματα. Μπορεί στο μέλλον άλλες ε, πανεπιστημιακές μελέτες μπορεί να έχουν άλλα αποτελέσματα. Τώρα για τη βιώσιμη ανάπτυξη βεβαίως και θέλουμε να συμβάλλουμε στο πρόγραμμα δράσης με ενθουσιασμό. Η συμβολή μας, ιδιαίτερα μέσω του ΛΑΜ, θα στοχεύει να προωθήσει τις βέλτιστες πρακτικές ούτω ώστε οι λύσει να προέρχονται από τι ίδιε τι αγορέ. Δηλαδή για τα θέματα τη υποβολής εκθέσεων και γνωστοποίηση ελπίζουμε να υπάρξουν κάποια πρότυπα μέσω προδιαγραφών, μέσω νομοθεσία, ούτω ώστε η αγορά να έχει την αναγκαία πληροφόρηση, ούτω ώστε να στραφούν περισσότερο οι χρηματοδοτήσει προ βιώσιμα προγράμματα. Και δεν πρέπει να αρκεστούμε στι ελάχιστε προδιαγραφέ. Μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερα. Η ΕΦΡΑΓ, όπου μπορεί να συμμετάσχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι από κάθε είδους προέλευση μπορεί να βοηθήσει πολύ σε αυτή την προσπάθεια. Ευχαριστώ πολύ ο Πρόεδρος. Δεν βλέπω να θέλει κανείς άλλο το λόγο. Μπορούμε να ολοκληρώσουμε αυτήν την τόσο καρποφόρα συζήτηση. Ευχαριστώ τον κύριο Ζων Πολ και τον κύριο Βότσμαν για την εργασία του για την μόνιμη συνεργασία και για την ε, δέσμευσή σας να λάβετε υπόψη και το ψήφισμά μας για το IFRS 17. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και Γκοζές. Πέρα από το ψήφισμα που φυσικά θα μελετήσουμε, θα σας πρότεινα όταν η Κομισιόν θα καθορίσει τον τρόπο λειτουργίας του ΛΑΜΠ, το οποίο θα βασιστεί στο, IFRS, στο, στο e συγγνώμη, τότε να τα ξαναπούμε με εσά, ούτω ώστε να συμβάλλετε περαιτέρω. Νομίζω πως θα ήταν σκόπιμο να συμμετάσχετε σε αυτή την πρωτοβουλία. Άριστα, ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Βεβαίως, προσβλέπουμε σε αυτό. Θα συνεργαστούμε για τα πιο πρακτικά θέματα και επί της ουσίας και επί της διαδικασίας και σας ευχαριστώ για αυτή την πρότασή σας. Ευχαριστώ πολύ. Η επόμενη συνεδρίαση είναι τη Δευτέρα 28 Μαΐου στις 7 στο Στρασβούργο. Κλείνει η συνεδρίαση. Ευχαριστώ πολύ.